So, first of all, let me... Καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Ξέρουμε όλοι γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διεξάγουμε την ακρόαση του προτινόμενου επιτρόπου ε, κυρίου Σμιτ, του αγαπητού μας συναδέλφου. Μπορεί να είναι καταπληκτική η συνεργασία μας μαζί του, αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τον εγκρίνουμε για να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε εδώ στην παρούσα ακρόαση. Καταρχάς θα ήθελα να θυμίσω ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το παράρτημα 7 του κανονισμού μας το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους προτινόμενους επιτρόπους με βάση την προσωπική τους ανεξαρτησία, την ευρωπαϊκή τους προσήλωση, τις ικανότητες και τα προσόντα, της γνώσης για το χαρτοφυλάκιο και τις επικοινωνιακές του ικανότητες και δεξιότητες. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω πριν από την ακρόαση ότι ο προτινόμενος επίτροπος απάντησε σε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο το οποίο κανονικά πρέπει να έχετε όλοι σας. Σύντομα θα ήθελα να σας εξηγήσω τη δομή της σημερινής συζήτησης. Ο προτινόμενος ε, επίτροπος θα κληθεί να κάνει μια εισαγωγική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει το 1 τέταρτο της ώρας. Επίσης θα έχει μέχρι 5 λεπτά στο τέλος της συνεδρίασης για κάποια καταληκτικά σχόλια. Μετά την εισαγωγή θα έχουμε χρόνο για 25 ερωτήσεις από όλους σας Uh, Η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα ε, με την αρχή του ping-pong, δηλαδή μέσα σε ένα πεντάλεπτο θα έχει ο ερωτών ένα λεπτό για την ερώτηση, ο προτινόμενος επίτροπος θα απαντά ε, για δύο λεπτά και το ίδιο βουλευτής μπορεί να κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση ενός λεπτού με ένα λεπτό απάντηση. Επειδή είναι πολλές ερωτήσεις και είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος, θα εξασφαλίζω με πολύ μεγάλη αυστηρότητα την τήρηση του χρόνου και παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας. Η Επιτροπή απασχόληση είναι η κύρια επιτροπή επιφορτισμένη με την παρούσα ακρόαση. Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων είναι συνδεδεμένη, καθώς και οι Επιτροπές Γυναικών και Πολιτισμού είναι προσκεκλημένες και καλωσορίζουμε τους συναδέλφους από τις άλλες Επιτροπές. Ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων ε, θα γίνει από τους συντονιστές των ε, πολιτικών ομάδων και ο δεύτερος γύρος βάσει ε, στη γενική κατανομή των ε, ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εκπροσώπων από, τις, από τους μη εγγεγραμμένους. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι έχουμε διερμηνία σε 23 γλώσσες. Όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα και πραγματικά σας καλώ να το κάνετε. Σας θυμίζω επίσης ότι αυτά που λέτε θα πρέπει να μεταφράζονται για να σας προλαβαίνουν λοιπόν οι διερμηνείς, να μην τρέχετε με υπερβολική ταχύτητα. Και ε, τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η συζήτηση θα μεταδίδεται απευθείας στο διαδίκτυο, στην ιστότοπο ε, του Κοινοβουλίου και επίσης ε, θα υπάρξει στην ίδια ιστοσελίδα και το βίντεο από την συνεδρίαση. Ο κύριος Σμιτ είναι γνωστό, σύντομη παρουσίαση του χαρτοφυλακίου είναι πάρα πολύ φιλόδοξο σύμφωνα με τα όσα μας παρουσίασε η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και θα ήθελα να τονίσω τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και την υλοποίησή του, καθώς επίσης και την εγγύηση για τα παιδιά που ελπίζω να προστατεύσει ε, τους πιο ευάλωτους πολίτες που είναι τα παιδιά μας. Ιδιαίτερα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και σε κοινότητες που είναι αποκλεισμένες ε, από την κοινωνία. Ως Σλοβάκα επιτρέψτε μου να εκφράσω την ισχυρή μου ελπίδα και πεποίθηση να αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης με έδρα την Πρατισλάβα, γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να συντονίζουμε τα κοινωνικά μας συστήματα, κοινωνικής ασφάλισης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σμιτ για 15 λεπτά. Madame la Présidente, Κυρία Πρόεδρε, κύριοι και κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα για αυτή την ακρόαση ενώπιόν σας. Ε, καταλαβαίνω την και συνειδητοποιώ την αποστολή που θα μου δοθεί αν την επιβεβαιώσει το Κοινοβούλιο. Να συνεργαστούμε μαζί. Η πολιτική και επαγγελματική καριέρα μου δείχνει ότι είμαι πεπισμένος για την ευρωπαϊκή διάσταση. Έχω λάβει μέρος σε μια σειρά δράσεων για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει πως η Ευρώπη θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις επόμενες γενιές να γνωρίζουν την ειρήνη, την ευημερία και την ελευθερία. Μιλάμε για αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα που θα μπορούν να ε, θα μπορούμε να βιώνουμε σε καθημερινή ε, βάση. Όπως λέει και η συνθήκη, πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των λαών. Πρέπει να έχουμε μία ανταγωνιστική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 3, όπως αναφέρθηκε και η εκλεγμένη πρόεδρος της Επιτροπής. Πρέπει να συμφιλιώσουμε το οικονομικό και το κοινωνικό πρέπει να ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική διάσταση. Αναφέρομαι στη δήλωση του Ζακ Τελόρ του 2016. Πρέπει οι ευρωπαϊκές ε, πολιτικές να μην θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική διάσταση, γιατί αλλιώς το εγχείρημα δεν θα πετύχει, δεν θα υποστηρίζουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ, υποστηρίζω αυτή την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη στους πολίτες. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης κάνει συγκεκριμένη την Ευρώπη που προστατεύει, που θωρακίζει τους πολίτες τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και απερίφραστα ενώπιόν σας δεσμεύομαι γι' αυτό. Δεσμεύομαι για το συντονισμό και τον διάλογο. Θα περάσω τώρα στα αγγλικά. Αν με επιβεβαιώσετε ως επίτροπο θα προσπαθήσω να πετύχω δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να ενισχύσω την απασχόληση, να προωθήσω μια, ένα εργατικό προσωπικό που θα έχει τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ψηφιακή μετάβαση. Θα είναι η εργασία στο κέντρο της δράσης μου, όπως και τα κοινωνικά δικαιώματα και η κοινωνική ένταξη. Η αγορά εργασία στην Ευρώπη είναι σημαντική. Πρέπει να προσαρμοστούμε προς τα πάνω, να προωθήσουμε τις συνθήκες διαφύωσης. Πρέπει η Ευρώπη να εγγυάται τις καλές ευκαιρίες και την πρόσβαση σε όλους, ειδικά στα άτομα με αναπηρία, στους μετανάστες, στους Ρωμά και στους πιο στερημένους. Θέλω να σπάσω τον κύκλο της φτώχειας που επηρεάζει τα παιδιά και να βελτιώσω την υποστήριξη προς τους νέους. Θα εργαστώ για να προωθήσω μια πιο δίκαιη Ευρώπη, μια βιώσιμη οικονομία, όπου τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν ένα κεντρικό ρόλο μαζί με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο που έχει προταθεί, τον Βάλτη Ντομπρόσκης, θα προσπαθήσω να ενισχύσω την κοινωνική διάσταση με βάση τον, κοινωνικό πυλώνα, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Στενά και τακτικά, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, του κοινωνικούς εταίρου και όλου του ενδιαφερόμενου φορεί, θα προσπαθήσω να προωθήσω και να επιδιώξω μια πιο δίκαιη και ε, Ευρώπη που συμπεριλαμβάνει τους πάντες είναι αυτή η κοινή πολιτική δέσμευση και των τριών θεσμικών οργάνων. Σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο θα φτιάξω ένα σχέδιο δράσης για να εφαρμόσω έναν πυλώνα και σε επίπεδο ενωσιακό και στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τα επιτέγματα του Προέδρου Γιούνκερ και τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ε, της εκλεγμένης Προέδρου Φοντερ Λάιεν. Ε, υπάρχουν πολλά εκατομμύρια πολίτες που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως νέοι. Φαίνεται ότι μειώνεται η ανεργία, αλλά όχι σε όλα τα κράτη-μέλη, όχι σε όλες τις περιφέρειες. Δεν αποφελούνται όλοι από αυτές τις θετικές εξελίξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά μας ε, μας ε, εξασφαλίζει δίκαιη αμοιβή και μια καλή διαβίωση πρέπει κάθε εργάτης στην Ένωση να έχει ένα ελάχιστο μισθό, ο οποίος θα είναι δίκαιος. Δεν είναι να έχουμε έναν ενιαίο μισθό παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επιδιώξουμε να φροντίσουμε να διατηρηθούν τα κοινωνικά μοντέλα των κρατών μελών. Θέλουμε όμως ισότητα στις ευκαιρίες. Θέλουμε οι άντρες και οι γυναίκες ε, να αισθάνονται ότι έχουν μέλλον αυτοί, τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους. Μέσα στα πλαίσια αυτών των προκλήσεων πρέπει να ενισχύσουμε και θα ενισχύσω την ε, εγγύηση για τους νέους και θα προωθήσω την εγγύηση για τα παιδιά. Η ισότητα των φύλων, η ισορροπία και είναι μέσα στις ε, προθέσεις μου. Θα προσπαθήσω να κλείσω το χάσμα της αμοιβή και το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και να εφαρμόσω την οδηγία για την εξισορρόπηση μεταξύ εργασιακού και ιδιωτικού βίου για τις άντρες και τις γυναίκες ταυτόχρονα. Ανησυχούμε λόγω της βάθυνσης των ανισοτήτων, λόγω της ανισότητας στα συστήματα αμοιβή και συντάξεων. Θέλουμε να έχουμε δίκαιου μισθού, η γύρανση να υποστηρίζεται, να υπάρχουν κοινωνικέ υπηρεσίε. Αυτά είναι σημαντικά για να πατάξουμε την ανεργία και να διασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη. Η κοινωνική οικονομία μπορεί εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο, ειδικά στι τοπικέ κοινωνίε, δημιουργώντα ε, κοινωνικό, μέρισμα. Ε, κάτι άλλο που εγώ ε, συγκεκριμένα επιδιώκω είναι η ασφάλεια στην εργασία. Δεν είναι αποδεκτό το 2019 άνθρωποι στην Ευρώπη ακόμα να κινδυνεύουν στο χώρο εργασίας τους. Θα προωθήσω την έγκριση περαιτέρω μέτρων για, ε, ε, ενάντια στα καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας. Πρέπει να σκεφτούμε περαιτέρω το θέμα της εργασιακής ασφάλειας και υγείας. Όταν είσαι επίτροπος ε, για την εργασία, είσαι επίσης επίτροπος για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της αγοράς μας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτέγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πολίτες της. Παρόλα αυτά, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν ότι αυτή η κινητικότητα ενέχει και κάποιες προκλήσεις, όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ. Ε, πρέπει να αντισταθούμε και να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις ευκαιρίες ε, και να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες ε, που ε, έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να κινηθούν εντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζοντας ε, τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης θα διασφαλίσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Θα υπάρχουν κοινέ επιθεωρήσεις. Από τη συζήτηση την περασμένη εβδομάδα σε αυτή την Επιτροπή γνωρίζω ότι η θέσπιση της Ευρωπαϊκής Αρχής Απασχόλησης είναι σημαντικό θέμα για όλους σας. Σας διασφαλίζω ότι γρήγορα θα συσταθεί και θα λάβει τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Οι προκλήσεις για την Ένωση είναι ο παγκοσμιοποιημένος κόσμος, το οικονομικό, το τεχνολογικό, το περιβαλλοντικό και το δημογραφικό στερέωμα. Οι άνθρωποι χρειάζονται συνοδεία, να μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να ενημερώνονται τις δεξιότητές τους όπως απαιτεί η οικονομία. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική για την καριέρα και τις δεξιότητες έτσι ώστε να συνοδεύεται η μετάβαση στην καριέρα του καθενός σε κάθε ηλικία. Θα διερευνήσω την ιδέα των μεμονωμένων ε, λογαριασμών μάθησης. Οι αγορές εργασίας ε, αλλάζουν λόγω της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει αποφασιστικά να δράσουμε για να περιορίσουμε τους κινδύνους, να διαμορφώσουμε τη μετάβαση και να δράξουμε τις ευκαιρίες. Είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη στο ψηφιακό μέλλον. Γι' αυτό χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενεργά να αντιμετωπίσουμε τις νέες μορφές επισφαλούς εργασίας. Θυμόμαστε όλη την οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές υφέσεις, να είμαστε σίγουροι ε, ότι η Ένωση θα μπορέσει να αντιδράσει με έναν κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο σε μελλοντικούς κλειδονισμούς. Η αντίσταση, το πόσο στεναρή είναι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση εξαρτάται από αυτό. Χρειάζεται ένα ε, σύστημα ασφάλισης το οποίο θα σχεδιαστεί σωστά και προσεκτικά για να έχει γρήγορη αντίδραση στα σοκ έτσι ώστε να ε, προστατεύει και ριζικά από την ανεργία. Η κοινωνική και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι δύο, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος η αξιοπρεπής εργασία, η ποιοτική εκπαίδευση, η ανισότητα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο αυτή τη στιγμή επανεπικεντρώνεται στους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει να έχουμε μια αξιοπρεπή εργασιακή ατζέντα για όλους. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τους συναδέλφους μου για να διασφαλίσω ότι τα διεθνή στάνταρ εργασίας ε, θα είναι στο κέντρο των εμπορικών συμφωνιών και των πολυμερών ε, διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλα αυτά ως επένδυση για το μέλλον. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, συν δηλαδή, είναι ένα εργαλείο που θα υποστηρίξει την εφαρμογή των αρχών ε, του πυλώνα δίνοντας τους πόρους. Η μετάβαση προς μία ε, ουδέτερη περιβαλλοντικά οικονομία ε, θα πρέπει να φτάσει σε όλους. Δεν πρέπει καμία χώρα, καμία περιφέρεια να μείνει πίσω. Με το ESF+, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα και με το Investing You και το νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα τα πετύχουμε αυτά εφόσον αυτά είναι στεναρά. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε και νέα νομοθεσία, η οποία θα εφαρμόζεται και θα μπαίνει σε ισχύ με σωστό τρόπο για να υπάρχει συντονισμός των πολιτικών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και να υπάρχει μια πιο απλή και λογική χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων, όπως και του κοινωνικού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών. Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει να προωθηθεί σε όλα τα επίπεδα και μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν βασίζεται σε ισχυρούς και αυτόνομους κοινωνικούς εταίρους. Οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να υποστηριχθούν επίσης, γιατί συνιστούν ένα θεμελιώδες τμήμα της της ε, οικονομίας της αγοράς. Ως Επίτροπος ε, θα εμπλακώ σε πλήρη διάλογο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο, αλλά και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους. Με αυτό το τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε την επιθυμητή ισορροπία, της αποτελεσματικές και αναλογικές πρωτοβουλίες ε, που θα σέβονται πλήρως την επικουρικότητα πιο πολύ από ποτέ ε, πρέπει να, η συζήτησή μας να βασίζεται στα γεγονότα. Εγώ θα βασίζομαι στην πλήρη ανάλυση, στην αξιολόγηση επιπτώσεων της κάθε πρωτοβουλίας που θα λαμβάνουμε. Θα αντλώ από την έμπνευση που υπάρχει και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους εταίρους μας στο G7 και στο G20, από τη συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς όπως το Ινδιεθή Οργάνωση Εργασίας και τον OECD. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η ε, εκλεγμένη πρόεδρος μας έδωσε ένα σαφές μήνυμα ως παρακαταθήκη. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να επιτύχει περισσότερα. Σήμερα ήρθε σε εσά με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Ο κατάλογος αυτός όμως δεν είναι εξαντλητικός, ούτε πλήρης. Θα πρέπει ε, σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς και γρήγορα εμείς να βρούμε το προσανατολισμό μας τις απόψει σα, τις ιδέες σας, τις ερωτήσεις, ακόμα και τι αντιρρήσεις σα, θα τι ακούσω και σα διαβεβαιώ ότι στην επόμενη πενταετία θα συνεργαστώ πάρα πολύ στενά με το κοινοβούλιο σα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των οικογενειών, των εργαζομένων και των εργοδοτών και να την ενισχύσουμε ξανά. Η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρος της υφηλίου για να ζει και να εργάζεται κανείς. Στόχος μου είναι να συνεισφέρω και εγώ προς την κατεύθυνση αυτή και ώστε να παραμείνει αυτό. Μαζί ε, θα πρέπει να διαμορφώσουμε τη δύναμη της Ευρώπης και την ισχύ της για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή ε, με όλο αυτό το ε, φιλόδοξο σχέδιο και ε, για τη τήρηση του χρόνου. Πριν δώσω το λόγο στους συντονιστές για τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η κυρία Αν Σαντέρ έχει γενέθλια. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. And now we'll Και τώρα θα περάσουμε στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Συντονιστέ των πολιτικών ομάδων. Γνωρίζετε το πεντάλεπτο και τις διαδικασίες, όπως σας είπα. Ο κύριος Ράτκε, λοιπόν, πρώτος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητέ συνάδελφε Σμιτ, αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι, η κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αρχή ε, που μας διέπει. Ορισμένοι εκπλήσονται ακόμα, παρόλο που είναι κατοχυρωμένα αυτά στη συνθήκη. Μήπως να διάβαζαν περισσότερη τη συνθήκη που είναι η βάση για τη δουλειά μας. Αλλά η κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι κοινωνική τότε μόνο ε, όταν λειτουργούν ε, στη συνεργασία τους οι κοινωνικοί εταίροι. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν λειτουργεί πλέον αυτό. Ε, από την άλλη βλέπουμε σε πολλά κράτη-μέλη ότι οι σχέσεις των κοινωνικών εταίρων είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο για τις κυβερνήσεις. Και τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ζήσαμε το γεγονός ότι αποκοιμήθηκε κάπου ο κοινωνικός διάλογος. Για μεταξύ άλλων, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ήμασταν αναγκασμένοι στην τελευταία θητεία ε, να κινήσουμε μια οδηγία για ε, τις ε, αξιόπιστες και σωστές συνθήκες και συνεννόηση στους χώρους εργασίας. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επόμενη πενταετία, πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, τον κοινωνικό διάλογο και πώς θέλετε να ενισχύσετε και να αναζωογονήσετε και πάλι την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συμφωνώ με την ανάλυση σας. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ε, βασίζεται στην ε, κοινωνική οικονομία της αγοράς και στον κοινωνικό διάλογο. Χωρίς ισχυρούς κοινωνικούς εταίρους και διάλογο φυσικά δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι η κοινωνική οικονομία της αγοράς όπως λειτουργούσε χρόνια ολόκληρα σε πολλά κράτη με μεγάλη επιτυχία και το τονίζω με μεγάλη επιτυχία και με στόχο να υπάρξει ευημερία για όλους. Ευημερία για όλους ήταν το σύνθημα σε μια μεγάλη χώρα, ε, από που το δημιούργησε και ο εμπνευστής της κοινωνικής οικονομίας αγοράς. Οι μεγάλες αλλαγές όμως ε, που οδήγησαν σε όλες τις χώρες και τα συνδικάτα των εργαζομένων και οι εργοδοτικές εργανώσεις αποδυναμώθηκαν. Και είναι πολύ σημαντικό σε ε, αυτές τις οικονομικές αναταράξεις να φροντίσουμε εκατέρωθεν οι κοινωνικοί εταίροι να ενισχυθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να το πράξει αυτό. Στην οικοδόμηση των θεσμών, όπως το λέμε σε αυτό το institution building, έχουμε πολλά μέσα και οικονομικά που θα πρέπει στοχευμένα να κινητοποιηθούν, ιδιαίτερα σε χώρες όπου ο κοινωνικός διάλογος είναι μάλλον άγνωστο, ξένη λέξη. υπολογίζω ε, και προσβλέπω πάρα πολύ και ποντάρω στον κοινωνικό διάλογο και θα πρέπει να καταλάβουν οι κοινωνικοί εταίροι ότι έχουν μέγα συμφέρον ε, να συνδιαμορφώνουν αυτό το κοινωνικό διάλογο και να πετυχαίνει αυτός. Γιατί συχνά η επιτυχία του ενός ταυτίζεται με την επιτυχία του άλλου. Η Ευρώπη είναι ε, μια τεράστια επιχείρηση, ένα εγχείρημα που προωθεί τον συμβιβασμό, τον επικοδομητικό όμως συμβιβασμό και η κοινωνική εταίρη και ο κοινωνικό διάλογος ζει από τους συμβιβασμούς. Αυτό ε, φέρει πιο κοντά την κοινωνία. Κύριο Ράτκε για συμπληρωματική ερώτηση. Ε, ε, εξαγγείλατε κάτι για κατώτατο μισθό, ότι στο προσεχές μέλλον θα το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για μένα είναι δεκανίκη ο κατώτατος μισθός. Τι θα πει αυτό, δίκαιος μισθός, σωστός μισθός, είναι αυτό που προκύπτει από τις συλλογικέ συμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται ε, να κάνει για να προωθήσει τις συλλογικέ συμβάσεις ε, που σήμερα έχουν υποχωρήσει. Είχα ένα συνάδελφο στο Λουξεμβούργο που έλεγε ε, ο κατώτατος μισθός είναι ο μισθός της συλλογική σύμβασης ε, για εκείνους που δεν έχουν συλλογική σύμβαση. Ε, γιατί δεν υπάρχει παντού αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη σε πολλές χώρες αποδυναμώθηκε πάρα πολύ και σε κάποιες άλλες σχεδόν έχει εξαφανιστεί, αποσιάζει τελείω. Αυτό έχει να κάνει με τον κοινωνικό διάλογο και εξαρτάται. Θα πρέπει να ενισχύσουμε πρώτα τους κοινωνικούς εταίρους και να τους δείξουμε ότι ο καλύτερος δρόμος είναι οι συλλογικές συμβάσεις, γιατί δίνει δικαιώματα σε όλους, αλλά και την ευελιξία που χρειαζόμαστε καμιά φορά στην οικονομία μας. Και όταν ε, ευημερεί ο κοινωνικός διάλογος σε μια καλή επιχείρηση, υπάρχει και αλληλοκατανόηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Αυτό πώς θα το καταφέρουμε. Ε, αυτό δεν ε, επιβάλλεται με ένα φυρμάνι, από αύριο όλοι θα υπογράψετε συλλογική σύμβαση. υπάρχει ο κοινωνικός διάλογος, αυτόν θα πρέπει να ενισχύσουμε και ε, να είμαστε ανοιχτοί και πάλι για τις συλλογικέ συμβάσεις και να πούμε ότι υπάρχει οικονομικό συμφέρον για τις συλλογικέ συμβάσεις. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να το σκεφτούμε. Με τον κοινωνικό διάλογο, αν υπάρχουν δρόμοι και τρόποι να τους αξιοποιήσουμε. Θέλω να τον αναθέσω αυτό στην ΟΚΕ. Να κάνει μια μελέτη η Ευρωπαϊκή Οικονομική ε, και Κοινωνική Επιτροπή για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πολιτική του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών συμβάσεων. Και ο ΩΣΑ εργάζεται ε, και ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας θα πρέπει να εμπνευστούμε. Η κυρία Γιονγκέριος. Thank you, President, Ευχαριστώ πολύ, ε, υποψήφιο επίτροπε Νίκολα Σμίτη για την εισήγησή σας. Είναι δίκαιο να πούμε νομίζω ότι η οικογένεια των σοσιαλιστών έχει αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Άρα δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι εμείς τονίζουμε και την εφαρμογή αυτού του πυλώνα. Ε, μιλήσατε για πρόγραμμα δράσης. Εγώ θα πρότεινα την αλλαγή του τίτλου σας Αντί για επίτροπο απασχόληση, να είναι επίτροπο ε, θέσεων απασχόληση και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η ερώτησή μου όμω είναι η εξή. Ποια θα είναι τα μέτρα και ποια θα είναι η οικονομική στήριξη που θα δώσετε έτσι ώστε η κοινωνική πρόοδο και η μετάβαση ηλικιακή προς μια ε, βιώσιμη κοινωνία να καταστούν πραγματικότητα για τους συμπολίτες μας. Δηλαδή όχι μόνο λόγια αλλά και πράξεις. Όταν υιοθετήθηκε ο κοινωνικό πυλώνα στο Γκέτεμποργκ, ορισμένοι ήμασταν κάπω προβληματισμένοι, γιατί λέγαμε αυτό, ότι άλλη μια δήλωση και μετά τι θα γίνει. Μετά όμω πολύ σύντομα διαπιστώσαμε πως υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερο δυναμικό σε αυτόν τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Υπό έναν όρο, ότι θα έχουμε την πολιτική βούληση να το εφαρμόσουμε, να το μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες ε, ενέργειες και δράσεις. Και αυτό σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή μας. Ε, Όμω αποτελεί αυτό και μια πρόσκληση ε, λόγω τη στρατηγικής ατζέντα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πολύ σύντομα λοιπόν, πολύ γοργά θα εργαστούμε επί αυτού του προγράμματος δράσης, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφράσουμε αυτές τις αρχές σε συγκεκριμένες δράσεις, σε ενέργειες. Μπορεί να είναι νομοθετικές πράξεις, μπορεί να είναι απλά συστάσεις, μπορεί να είναι ιδέες που τα κρατημέλη θα χρειαστεί να μεταφράσουν στην πράξη γιατί θα πρέπει να σεβαστούμε τις αρμοδιότητες των κρατών μελών και τις αρμοδιότητες της Ένωσης, που συχνά είναι και κοινέ. Ήδη μέσα στην επιστολή της εντολής μου ε, υπάρχουν κάποια πράγματα που δηλώνονται ρητά. Ελάχιστος μισθός, ε, εγγύηση για τα, παιδιά. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε τι εννοούμε. Έχουμε και την εγγύηση για την νεότητα θα πρέπει αυτή να την αναβαθμίσουμε γιατί οι νέοι χωρίς δουλειά, οι νέοι άνεργοι είναι το χειρότερο για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Πρέπει να ενθαρρύνουμε λοιπόν, την την... να ενισχύσουμε μάλλον την εγγύηση για τους νέους να δούμε με ποιον, ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να εφαρμόσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα και τις καλές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες αυτά είναι κάποια ε, κάποιες άξονες όπου χρειάζεται να έχουμε νομικά μέσα στη διάθεσή μας και τώρα για τα οικονομικά θα πρέπει το κοινωνικό ταμείο να συμβάλλει στην εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα φυσικά. Κυρία Γιουγκέριους, έχετε συμπληρωματική ερώτηση μάλιστα και αυτή εστιάζεται στην εγγύηση για τα παιδιά. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσφαση, τη δέσμευση της Κομισιόν ως προς, αυτόν, ε, ε, ως προς αυτό. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρίσκεται στην ατζέντα της Κομισιόν. Ερώτησή μου όμως είναι τι είδους μέσο και τι είδους χρηματοδότηση προβλέπει η Κομισιόν για αυτή την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά. Και πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη να στηρίξει αυτή την πρόταση να στηρίξουν αυτή την πρόταση στις διαπραγματεύσεις και να δώσουν φρέσκο χρήμα αντί να, να, ε, να μετακινήσουν μάλλον χρήματα από άλλους τομείς ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλοι συμφωνούμε ότι η παιδική ένδια είναι αυτή που καταστρέφει το μέλλον των ε, φτωχών παιδιών. Το να είναι κανείς φτωχό παιδί σημαίνει πως θα είναι συνήθως και φτωχό ενήλικας. Είναι φρικτό για το άτομο, αλλά είναι φρικτό και για την κοινωνία. Ήδη τώρα υπάρχουν πολλά μέσα και μέτρα που λειτουργούν για τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών. Πρέπει όμως αυτά όλα να τα συγκεντρώσουμε και να τα συνδυάσουμε πρώτα απ' όλα για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο μέσα στην κοινωνία μας. Και θα πω ότι δεν είναι μόνο για την κοινωνία, αλλά ε, ε, για τις στοχές κοινωνίες, αλλά και στις πλούσιες κοινωνίες έχουμε φτωχά παιδιά και θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και μπορώ να φανταστώ με βάση τη δουλειά που έχει γίνει στο Κοινοβούλιο να κάνουμε κάποιες συστάσεις. Τα χρήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε φιλόδοξη πολιτική που να είναι καλή για όλου και θετική χωρί να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Εγώ σημειώνω τα όσα λέει το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπο που σκεφτήκατε και βεβαίω θα το φέρω σε συζήτηση και με το Συμβούλιο. Μάλιστα. Πισλάρου, ένα λεπτό. Ε, ερώτηση. αυτό το χαρτοφυλάκιο χρειαζόμαστε ένα μαχητή, έναν αγωνιστή για να ενισχύσουμε και το status quo. Οι πολίτες στις 26 Μαΐου μας έδειξαν ότι ελπίζουν στην Ευρώπη. Και η ομάδα μας, το Renew Europe, εκπροσωπεί αυτή την αναγέννηση για να ανταποκριθούμε στα όνειρα και τις προσδοκίες ε, των ε, πολιτών. Ξέρω πόσο έμπειρος είστε και είμαι βέβαιος ότι θα είστε και φιλόδοξος επίτροπος για να προωθήσετε αυτά τα θέματα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε σε δεινή κατάσταση. Έχουμε πάνω από 25% των παιδιών μας να ζουν στη φτώχεια και είναι περιορισμένες ε, οι ευκαιρίες για τους νέους. Ε, έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, έχουμε την εγγύηση για την νεολαία ε, και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα για την νεολαία. Πώς σκοπεύετε να συνδέσετε ε, ε, την εγγύηση για την νεολαία με την μελλοντική ατζέντα για την απασχόληση αυτού του θεματολόγιου. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω και το είπα προηγουμένως για την εγγύηση για την νεολαία, θα πρέπει να επανεφεύρουμε, να προσαρμόσουμε αυτή την εγγύηση στην παρούσα κατάσταση. Έχει πετύχει πολύ αυτό το πρόγραμμα, όχι παντού με τον ίδιο τρόπο, αλλά γενικά έχει πετύχει. Τώρα όμως αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Πρώτον, έχουμε το ζήτημα ε, της επισφάλειας των νέων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας με πολύ επισφαλείς συνθήκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει οπωσδήποτε και να ασχοληθούμε. Ε, γιατί θα πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στους νέους να χτίζουν τη ζωή τους σε πιο γερά θεμέλια, μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεύτερον, η κατάσταση της ψηφιακής μετάβασης ε, κυριαρχεί παντού. Ακόμα και οι νέοι, παρόλο που όλη την ώρα παίζουν με τα κινητά τους τηλέφωνα, δεν έχουν πάντα τα εφόδια εκείνα και τη γνώση για να μπουν σε αυτή τη νέα ψηφιακή εποχή. Και μία από τις ιδέες μου θα είναι να εισαγούμε για κάθε νέο, μέσω της εγγύης νεολαίας ή για κάθε νέο άνεργο, ένα, ε, ε, μια βασική εκπαίδευση θεμελιώδη ε, για τα ψηφιακά ζητήματα, ανάλογα με τη γνώση του, με τη θέση την οποία φιλοδοξεί να καταλάβει για να έχει ε, ε, τα εργαλεία όλα και τα εφόδια να μπει στην ψηφιακή αγορά. Μια βασική κατάρτιση. Θα ζητήσω από τη Γενική μου Διεύθυνση λοιπόν πώς θα δώσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες στους νέους. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και με τους άλλους επιτρόπους ε, που είναι αρμόδιοι για ψηφιακά θέματα, για την παιδεία. Πώς μπορούμε πραγματικά να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, να δώσουμε μια όθηση στους νέους για να μπουν στην ψηφιακή αγορά και στην ψηφιακή κοινωνία. Για να υπάρχει και μια καλή ευκαιρία για αυτούς και όχι μια, ε, μια περίοδος αβεβαιότητας και πολλών κινδύνων. Έχετε την επερώτησή σας κύριε Πίσα. Πολύ τολμηρό και φιλόδοξο αυτό που σχεδιάζετε. Θα δημιουργήσετε μια νέα μονάδα ε, στην ε, Γενική σας Διεύθυνση ακόμα και Διεύθυνση για την νεολαία. Και ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια για να δημιουργήσετε αυτή τη δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης με μια διαβίου μάθηση ας πούμε και μετεκπαίδευση ε, Ας πούμε υπάρχουν προβλήματα ψηφιακά ε, που αφορούν τους μηχανικούς, που αφορούν ε, τους υδραυλικούς, ε, που αφορούν τους ξυλουργούς. Έχουν μπει τα ψηφιακά και εκεί ας πούμε και στα υδραυλικά και σε όλα αυτά. Ε, ακριβώς πολύ ωραία το είπατε. Χρειάζεται καλό συντονισμό, το είπα και εγώ προηγουμένως, μεταξύ των διαφόρων επιτρόπων και θα πρέπει να οργανώσει και ο Αντιπρόεδρος ε, αυτά τα θέματα. Εγώ έχω διατελέσει υπουργό Απασχόλησης και πάντα εργάζομαι στενά με τους διάφορους επιτρόπους ε, και ε, με τον Επίτροπο Σχοινά. Η επαγγελματική κατάρτιση Ε, η επαγγελματική κατάρτιση δεν είναι η δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, επειδή δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο, καλά πας στην τεχνική εκπαίδευση. Όχι. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ε, κορυφαία και εξίσου με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ η Επιτροπή σας έχει προωθήσει πολύ ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο την ε, επαγγελματική κατάρτιση και πέραν αυτών. Και οι πάντες γνωρίζουν ότι εκεί που είναι ισχυρή η επαγγελματική κατάρτιση η ενεργεία των νέων είναι χαμηλή. Και αυτή είναι η βάση στην οποία θα πρέπει να οικοδομήσουμε. Και εκεί θα πρέπει να ενταχθεί η ψηφιακή λογική και με νέε μεθόδους κατάρτισης. Πέρα από τα γνωστά πλαίσια και τα κλασικά του εκπαιδευτικού συστήματος. I'm speak in Danish to avoid any misunderstanding. Θα μιλήσω δανέζικα για να μην υπάρχουν ε, κάποιες παρεξηγήσεις. Ε, είμαστε σε μια εποχή όπου βιώνουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουμε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής μέσα σε αυτή την αλλαγή. Η δική μου γενιά και οι φίλοι των Παρασκευών για το μέλλον θέλουμε να ε, αγκαλιάσουμε αυτή την αλλαγή για να έχουμε μια δίκαιη μετάμβαση, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να έχουν μια βάση στη ζωή τους, να μην πέσουν στη φτώχεια, να έχουν ευκαιρίες για τους αγαπημένους τους. Στη Δανία έχουμε μάθει ότι το υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας ενισχύει τους εργαζομένους ε, στο να ε, αγκαλιάσουν τη διαβίου μάθηση. Θα προωθήσετε ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο εισόδημα, δεν είναι το ίδιο με τον ελάχιστο μισθό, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι να είναι πιο ευέλικτοι και να μπορούν να προσαρμοστούν χωρίς ε, να φοβούνται ότι θα πέσουν στη φτώχεια. Η απάντησή σας, δύο λεπτά. Καταρχάς, να πω ότι αυτό που αναφέρατε στην αρχή είναι κοινή ανησυχία. Χρειαζόμαστε να διαβάσουμε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ε, της εκλεγμένης Πρόεδρου της Κομισιόν. Θέλουμε μια Ευρώπη ε, κοινωνική, κοινωνικής ευημερίας, δικαιοσύνης και αυτό πρέπει να επιδιώξουμε, γιατί ακριβώς η ιστορική εμπειρία αυτό δείχνει ότι Κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εγγυημένο. Ακόμα και οι Ευρωπαίοι μπορεί να τρελαθούν, πολιτικά να τρελαθούν. Αυτό είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού όμως, ε, τρόπου ζωής, ε, στην κοινωνική αγορά. Τώρα για το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα. Στις περισσότερες χώρες, νομίζω σχεδόν σε κάθε χώρα, σε κάθε κράτος μέλος, έχουμε κάποιο είδους ελάχιστο εισόδημα. Αλλά αυτό τα διαφέρουν. Κάποια είναι σε χαμηλά σε επίπεδο ποσών, άλλα πολύ ψηλά. Μπορεί να μου πείτε ότι υπάρχει επικουρικότητα. Όχι, υπάρχει και κάτι κοινό, κοινό συμφέρον στο να εγγυηθούμε ότι ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Ακόμα και αν αυτό το άτομο αύριο δεν μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας αύριο και να βγάλει τα προστοζήν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε κάποιου είδους κριτήρια, κάποιους συγκρίσιμους όρους για να μπορεί ο κόσμος να ζει αξιοπρεπώς. Όπως είναι και ο ελάχιστος μισθός, έτσι είναι και το ελάχιστο εισόδημα στο Λουξεμβούργο, στη Βουλγαρία ή οπουδήποτε αλλού. Ό,τι και να είναι πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι συνολικά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένο βιωτικό επίπεδο. Υπάρχει μια οικονομική, χρηματοπιστωτική κατάσταση και πρέπει να εγγυάται σε κάθε πολίτη, όπου και αν βρίσκεται στην Ευρώπη, μια αξιοπρεπή διαβίωση. Επί αυτού πρέπει να επικεντρωθούμε και να εργαστούμε. Και αυτό πρέπει να γίνει με μια κατάλληλη μελέτη με συζήτηση, διάλογο με τα κράτη-μέλη και φυσικά με όλους τους οργανισμούς που ασχολούνται με την ανέχεια και τη συμπερίληψη. Θέλω πραγματικά να ακούσω τι έχουν να μου πούν η επερώτηση. Ευχαριστώ πολύ καλό που το ακούω αυτό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα αναλάβετε την υποχρέωση ε, να συζητήσετε το θέμα αυτό με τους ε, αντιπροέδρους Τίμερμανς και Ντομπρόφσκης για να, στις πρώτες 100 μέρες ε, για να έχουμε μια γρήγορη μετάβαση. Συγγνώμη, άρχισε αργά η μετάφραση και δεν κατάλαβα την ερώτηση. Χαίρομαι για την απάντησή σας. Θέλετε αυτή το θέμα να το θέσετε στους ε, αντιπροέδρους Τίμερμανς και Ντομπρόφσκης για να περάσει αυτό στο πρόγραμμά σας στις πρώτες 100 μέρες. Δεν μπορούμε να τελειώσουμε τη δουλειά στις πρώτες 100 μέρες, γιατί δεν θα έχουμε τι να κάνουμε στην υπόλοιπη μας. Όμως, είναι ξεκάθαρο πως ο κόσμος περιμένει από μας ένα μήνυμα, γρήγορα και ξεκάθαρα. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι τα καλύτερα εργαλεία ή τα καλύτερα μέσα. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την πρόθεση αυτών των στάνταρτ. Αυτό θα γίνει γρήγορα, δεν θα αρχίσουμε στο τέλος της θητείας, θα το κάνουμε άμεσα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι χρειάζεται διαβούλευση, επιμένω πολύ στη διαβούλευση, γιατί εμείς οι επίτροποι δεν τα ξέρουμε όλα, υποθέτω. Πρέπει λοιπόν να διαβουλευτούμε με αυτούς που κάποιες φορές ξέρουν περισσότερα από εμά. Η κυρία Ζαμέ. Κύριε Πέτροπε, ε, τα θέματα τα κοινωνικά και απασχόληση είναι αυτά που απασχολούν περισσότερο του πολίτες μας. Υπάρχουν προκλήσεις και κίνδυνοι. Υπάρχουν νέε χώρε ε, που έχουν βασιστεί στην υπερκατανάλωση και την, ε, το ατελείωτο κέρδο που μα οδηγούν ε, σε, στα προβλήματα που γνωρίζουμε. Η ευρωπαϊκή πολιτική λιτότητα επηρεάζει τι συντάξει. Η ευρωπαϊκή πολιτική ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασία περιορίζει τι επιλογέ των ετούντων εργασία έχουμε καταλήξει στη μείωση των δικαιωμάτων, στην περιορισμό των δικαιωμάτων και με το κοινωνικό dumping που οργανώνεται γύρω από την αποσπασμένη εργασία, τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ερώτηση, πότε θα αφήσετε την οικονομία να εξυπηρετεί τους ανθρώπους και όχι το αντίστροφο και έπειτα πότε θα μπούμε εμείς στην υπηρεσία των λαών και όχι το αντίθετο η υποψήφια πρόεδρος έχει ορίσει ένα ε, ε, στόχο να τοποθετήσουμε όχι μόνο την Ένωση αλλά και την οικονομία στην υπηρεσία ανδρών και γυναικών. Και όλα όσα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της και όσες είναι οι, κεντρικοί, οι κεντρικές γραμμές, οι κεντρικοί άξονες τους οποίους σας εξέθεσα έχουν ένα στόχο, να ενισχύσουν την κοινωνική προστασία, την κατάσταση της κοινωνικής προστασίας στην Ευρώπη, να ενισχύσουν και να ε, τονώσουν ε, το κοινωνική πρόοδο με προσαρμογή σε μια οικονομία που αλλάζει, σε ένα κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει, δηλαδή και η παγκοσμιοποίηση. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε αγαθοί ε, σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει εκεί να συμβάλλουμε, να συμβάλλουμε με τις ιδέες και τις αντιλήψεις μας ε, στη διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. Για το κοινωνικό ντάμπινγκ πιστεύω πως η Κομισιόν έχει κάνει προτάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την απόσπαση εργαζομένων που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί διότι ακόμα είμαστε σε φάση μεταγραφής της οδηγίας αλλά η αρχή που είναι βασική αρχή και που θα πρέπει να την, προσέξουμε και πρέπει οπωσδήποτε να την εφαρμόσουμε είναι ο ίδιος μισθός γιατί στο για την ίδια εργασία σε οποιοδήποτε ε, μέρος. Αυτό είναι μια μικρή επανάσταση και όταν ξεκινήσαμε με την, με την οδηγία περί αποσπασμένων εργαζομένων δεν ήταν κάτι το δεδομένο αυτό, όμως το έχουμε καταφέρει και θα συνεχίσουμε ε, να επιμένουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική προστασία, πρόνοια με το μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας, που είναι οι συστάσεις για την κοινωνική προστασία όλων και την ένταξη όλων. Και γι' αυτό μιλάμε για εγγύηση για τα παιδιά, για τους νέους. Όλα αυτά στόχο έχουν να ενισχύσουν το κοινωνικό κράτος για το οποίο η Ευρώπη να είναι περήφανη. Επερώτηση. Υπερώτηση της κυρία Ζαμέ. Ναι, θέλω μια διευκρίνηση. Η ουμπεροποίηση δεν είναι ε, κάτι το αποδεκτό για την κοινωνία μας. Θα, το, συμφωνείτε φαντάζομαι. Σε μένα, στη δική μου περιφέρεια ε, εξαφανίζονται οι μαθητευόμενοι γιατί καλούνται οι μετανάστες. Ε, εξαφανίζονται διάφορα επαγγέλματα. Εγώ βρίσκω ότι σε αυτή την αρμόνιση των μισθών ε, μιλάμε για μία μείωση προς τα κάτω. Νομίζω πως ε, το ξέρουμε όλοι αυτό και εσείς οι ίδιοι όταν μιλάτε και ανακοινώνετε μελλοντικέ κρίσεις και διευκρινίζετε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, έχουμε, να καταφέρουμε να έχουμε τη στήριξη των συμπολιτών που δεν την έχουμε τώρα, ε, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αναφέραμε την προστασία των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Αυτό που λέτε ουμπεροποίηση είναι ταυτοπροσωπία. Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα εργαστεί πάνω στην προστασία της συνθήκες εργασίας Τη κοινωνική προστασία και πρόνοιας των εργαζομένων στις πλατφόρμες. Αυτός είναι ένας σπουδαίο στόχο και είναι κάτι που ε, πρέπει πολύ γρήγορα να ε, αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει στις 100 μέρες, αλλά πάντως σίγουρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι μια οικονομία που επεκτείνεται και αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία και δεν έχει μόνο άρχισιμες πτυχές και όπου σίγουρα υπάρχει ανάγκη να ε, εισαχθεί κοινωνική ρύθμιση. Ε, δηλαδή η κοινωνική πρόνοια δεν μπορεί να σέρνεται πίσω από την τεχνολογική εξέλιξη. Ε, το είπαμε αυτό και θέλουμε να, να επενδύσουμε, λέει. Ακούω διάφορες φωνές που έρχονται και από άλλες χώρες και από, αυτές, και από τη δική σας ώρα, ότι έχουμε, θέλουμε να επενδύσουμε στην κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση των νέων και στην δυτή αυτή κατάρτιση ε, μαθητεία και κατάρτιση. Δηλαδή να βρούμε, να μπεκεδεύσουμε τους νέους ώστε να μπορούν να βρουν δουλειά και με την απαραίτητη κοινωνική προστασία. Ευχαριστούμε. Κυρία Ραφάλσκα, ένα λεπτό για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την κινητικότητα των εργαζομένων. Αυτά είναι πολύτιμα. Αλλά αυτή τη στιγμή η δουλειά που γίνεται αφορά την αναθεώρηση ε, των νομοθετημάτων. 987 και 893 για τη μείωση ε, των εμποδίων που γνωρίζουν οι ε, εργαζόμενοι, αλλά τώρα αυξάνεται η γραφειοκρατία αντί να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι. Οι διεθνείς μεταφορές ή ο τομέας της υγείας ε, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω αν προτίθεστε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Είναι πολλές οι χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, ε, που προτίθενται να απορρίψουν τις νέες σας ε, ιδέες και προτάσεις. Συμφωνώ απολύτως όταν λέτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύτιμες και για την οικονομία μας και για την ανάπτυξή μας και για τις θέσεις απασχόλησης και εργασίας. Είναι εκείνες οι εταιρείε που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Είτε δουλεύουν σε μεγάλη εταιρεία είτε σε μικρομεσαία. Κάθε πολίτης, κάθε εργαζόμενος στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να έχει ένα αξιοπρεπή μισθό και σωστέ συνθήκε εργασίας. Θα πρέπει να βοηθούμε, να υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε αυτές τις αλλαγέ που είναι υποχρεωμένε να κάνουν και είναι προφανέ. Θα πρέπει να τις ε, οχυρώσουμε για τη νέα ψηφιακή οικονομία, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούμε να χτίσουμε τις μελλοντικές μικρομεσαίες σε κακά θεμέλια, σε πολύ χαμηλούς μισθούς και κακές συνθήκες εργασίας. Δεν είναι αυτό το μέλλον του οικονομικού μοντέλου στην Ευρώπη. Συμφωνώ ότι το ζήτημα του διοικητικού ε, άχθους ε, παραμένει υψηλή προτεραιότητα για μας. Θα πρέπει να ελέγχουμε αυτά τα εμπόδια, να μην καταστρέφουν την ανταγωνιστικότητα ε, των ε, μικρομεσαίων. Γι' αυτό είπε και η Πρόεδρος ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή κάθε φορά που προχωρούμε σε νέα νομοθεσία. Θα πρέπει να εκτιμούμε και να αξιολογούμε αν χρειάζεται αυτή η νέα νομοθεσία. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται οικονομία κάποιο είδους πλαίσιο κανονιστικό. Και στο, στην 883, 883 υπάρχουν διευκολύνσεις εγώ ε, εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη νέα μας ψηφιακή δυνατότητα να γίνουν τα πράγματα πιο διαφανή και πιο εύκολα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες. Ιδιαίτερα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ανταλλαγών Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου πολύ ε, γρήγορα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες τα συστήματα και τα ταμεία και να υπάρχει ε, μια κοινωνική ταυτότητα, δελτίο ταυτότητας για τους εργαζομένους. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική ε, που μου λείπει λίγο, είναι και η οικογενειακή πολιτική. Πολύ λίγος λόγος γίνεται για την οικογένεια. Και εγώ θεωρώ ότι βάλετε η οικογένεια, καταστρέφεται, ε, επανορίζεται στην Ευρώπη. Ποιο είναι ο ρόλο που βλέπετε για την οικογένεια στην ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι η οικογενειακή πολιτική είναι αυτόνομη, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνικούς στόχους χωρίς να σκεφτόμαστε την οικογένεια. Στην Πολωνία υπάρχει και παροιμία που λέει ισχυρή οικογένεια σημαίνει ισχυρή Πολωνία. Για την υπόλοιπη Ευρώπη αυτό βρίσκει εφαρμογή και μετάφραση. Συμφωνούμε όλοι ε, ότι η κοινωνία είναι ε, θεμελιώδης για η ε, οικογένεια για την κοινωνία μας. Κανείς δεν τον αμφισβητεί αυτό. Όταν μιλούμε για εξισορρόπηση του εργασιακού με τον ιδιωτικό βίο, όταν μιλούμε για πάταξη της ένδυας με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να βοηθούμε, να υποστηρίζουμε, να ενισχύουμε τις οικογένειες. Γιατί η παιδική ένδυα, πρώτα απ' όλα είναι οικογενειακή ένδυα. Τα φτωχά παιδιά ζουν σε φτωχέ οικογένειε. Γι' αυτό θα πρέπει να χαράξουμε πολιτικές, όχι μόνο για τα παιδιά, για να βοηθήσουμε και τις οικογένειε. Δεν καταλαβαίνω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να βοηθάει και να υποστηρίζει τις οικογένειε. Το κοινωνικό μας μοντέλο ακριβώς αυτό κάνει. Ενισχύει και βοηθάει τι οικογένειε, δίνοντα τους καλές κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες και τη δυνατότητα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να έχουν μια καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πραγματικά ίσες ευκαιρίες. Family which... Και ε, αυτή είναι πραγματικά η ενεργή οικογενειακή πολιτική που εμείς υποστηρίζουμε. Αλλά ε, συμφωνώ, είναι κυρίως ε, εθνική αρμοδιότητα οι πολιτικές για την οικογένεια, αλλά θα πρέπει να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες και τις βασικές αρχές για τις μη διακρίσεις. Παρακαλώ οι επερωτήσεις θα πρέπει να έχουν πάντα να κάνουν με την αρχική ερώτηση. Ε, ο κύριος Βίλουμσεν. Στο Πρόεδρε θα μιλήσω δανέζικα. Κύριε Σμιτ, στην γραπτή απάντησή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον Ελάχιστο Μισθό θα πρέπει να σέβεται τις αρμοδιότητες των κρατών μελών αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους και τις εθνικές παραδόσεις σχετικά με τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ε, κατά πόσο θα εγγυηθείτε ότι ο ελάχιστος μισθός ε, που θα θεσπιστεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα σεβαστεί τις χώρες που δεν έχουν ελάχιστο μισθό αλλά ε, δια, διασφαλίζουν όπως εμείς κάνουμε στις βόρειες χώρες έναν ελάχιστο μισθό μέσω των συλλογικών συμβάσεων. Πώς ακριβώς θα το διασφαλίσετε αυτό μπορείτε να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Μιλήσαμε για τη σημασία, για την ε, ουσιώδη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πώς ε, θα υποστηρίξουμε, θα αναπτύξουμε, θα ενισχύσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλη την Ευρώπη. Πώς εγώ λοιπόν όταν έχω πει κάτι τέτοιο, όταν συμμερίζομαι αυτή την άποψη, πώς μπορώ να εξασθενήσω ένα σύστημα που βασίζεται στις συλλογικές συμβάσεις και που έχει δράσει τόσο επιτυχημένα ως τώρα γιατί ε, έχει καταφέρει να θεσπίσει καλούς μισθούς ε, και δικαιοσύνη στο χώρο της εργασίας. Αυτό το πλαίσιο για την ελάχιστη αμοιβή σε καμία περίπτωση, και αυτό το τονίζω, σε καμία περίπτωση δεν θα αμφισβητήσει το σύστημα ε, που βασίζεται στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις και διασφαλίζει καλούς μισθούς στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποχρεώσουμε αυτές τις χώρες να αλλάξουν μια παλιά και καλά παγιωμένη παράδοση. Και παρεπιπτόντως δεν έχουμε και την πρόθεση να φτιάξουμε έναν ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό. Πώς θα μπορούσαμε. Αυτό που θέλουμε είναι να φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Ειδικά στις χώρες που αυτό το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν υφίσταται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι θεσπίζονται ελάχιστες αμοιβέ με έναν διαφανή και προβλέψιμο τρόπο. Αυτό είναι το πλαίσιο που πρέπει να θεσπίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πειράξουμε την παράδοση και την κουλτούρα των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες όπου οι μισθοί και οι ελάχιστοι μισθοί προκύπτουν από κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ένα τέτοιο σύστημα. Θέλουμε να το διασφαλίσουμε, να το διατηρήσουμε και θα έλεγα σε πολλές χώρες να το αντιγράψουν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, κύριε Βίλουμσεν. Ευχαριστώ, κύριε Σμιτ. Ως επερώτηση. Μπορείτε παρακαλώ να μου απαντήσετε εάν συμφωνείτε ότι η νομοθετική πρόταση για την ελάχιστη αμοιβή θα πρέπει να περιλαμβάνει μια εξαίρεση λοιπόν για αυτές τις χώρες που έχουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όπου η ε, αγορά εργασίας καλύπτεται από τις συλλογικέ ε, διαπραγματεύσεις και τις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας. Αν θέλετε να το πείτε εξαίρεση, πείτε το έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Το είπα ξεκάθαρα δεν θα αλλάξουμε, δεν θα ενοχλήσουμε αυτό το σύστημα, ούτε θα του δημιουργήσουμε προβλήματα μέσα από αυτό το πλαίσιο για την ελάχιστη αμοιβή που θέλουμε να φτιάξουμε. Θα διατηρήσουμε ότι λειτουργεί καλά. Δεν επιδιορθώνεις κάτι που λειτουργεί καλά. Αυτή είναι η εγγύηση που μπορώ να σας δώσω. Δεύτερος ε, γύρος ε, ερωτήσεων. Είμαστε ήδη ε, δέκα λεπτά καθυστερημένοι. Γι' αυτό παρακαλώ να είστε πολύ ακριβείς. Ξεκινάμε με την κυρία Φράνσεν το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η ψηφιακή ανάπτυξη και η ανάπτυξη της οικονομίας των πλατφορμών ε, δίνει μεγάλες ευκαιρίες και για τους εργαζομένους ε, και για τους αυτοπασχολούμενους και είναι καλό. Από την άλλη αυτή η οικονομία όμως έχει και κάποια αρνητικά στοιχεία. τα ακούσαμε για, για τις ε, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις βραχυχρόνιες, τη μερική απασχόληση κτλ. Ε, ρωτώ, ε, η κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους πώς θα είναι εγγυημένη και είστε πρόθυμοι ε, του σημερινούς ε, ε, κανόνες και την ομοθεσία, όπως είναι η αποσπάση των εργαζομένων να την επεκτείνεται και στην ψηφιακή οικονομία και στις πλατφόρμες έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας αυτών των εργαζομένων. As um, Όπως είπα προηγουμένως, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις um, δεν θα μας ξεφύγουν γιατί η κοινωνική προστασία και οι κοινωνικές εγγυήσεις που έχουμε δημιουργήσει στην Ευρώπη τελικά ε, να μην καταστραφούν από αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Όπως ίσως γνωρίζετε, στις Ηνωμένε Πολιτείες, στην Καλιφόρνια παρακαλώ, τώρα έχουν περάσει νομοθεσία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εκεί γεννήθηκε και εφευρέθηκε όλη αυτή η οικονομία των πλατφορμών και έχουν καταλάβει ότι υπάρχει έλλειμμα και χάσμα ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες και την τεχνολογική ανάπτυξη. Και αυτό το έλλειμμα πρέπει εμείς να καλύψουμε. Τι έχει αρχίσει ήδη να κάνει η Επιτροπή αυτή με την οδηγία ε, για τις προβλέψιμες και διαφανείς συνθήκες εργασίας. Η Επιτροπή Απασχόλησης του Κοινοβουλίου δηλαδή, ε, με την κοινωνική προστασία που ε, καλύπτει και τους αυτοαπασχολούμενους, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ενισχύονται και αναπτύσσονται αυτά τα δικαιώματά τους. Ότι οι άνθρωποι αυτοί που εργάζονται σε πλατφόρμες έχουν τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με όλους τους άλλους εργαζομένους. Και θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα, ναι, και στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις κατά τα άλλα και συμβάσεις. Δηλαδή, ε, να μπορούν να συνεργάζονται και αυτοί με τις πλατφόρμες και που θεωρούνται αυτοπασχολούμενοι να μην έχουν, να ε, ε, εμπίπτουν μάλλον στο δίκαιο του ανταγωνισμού αλλά να έχουν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μια συνολική προσέγγιση λοιπόν για τις κοινωνικές ε, συνθήκες και εργασιακές συνθήκες και των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Το θα πρέπει να το συζητήσω με την κυρία Βεστάγκερ αλλά και τον Επίτροπο ε, της Βιομηχανίας και πολύ γρήγορα θέλω να διοργανώσω μια μεγάλη διάσκεψη με όλους τους ενεχομένους, τους ενδιαφερομένους και να αναπτύξουμε καλές ε, προδιαγραφές και πρότυπα για αυτή τη νέα ψηφιακή οικονομία. Ε, κυρία Φράνσεν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, κανείς δεν θα με παρεξηγήσει που ως Βελγίδα θέλω να σας πω ότι έχουμε να αποθέσει μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες στο πρόσωπό σας για να συνεχίσετε την καλή δουλειά που έκανε η προκάτοχό σας, η Μαριάν Τέισεν. Ε, και μια δεύτερη ερώτηση. Ε, τι γίνεται με τους ψευδό αυτοαπασχολούμενους. Αναφερθήκατε λίγο σε αυτό. Ε, το θέμα αυτό εκρεμεί εδώ και καιρό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα των αυτοπασχολουμένων. Well, no... Κοιτάξτε, κανείς δεν θέλει να επιτεθεί στους αυτοπασχολούμενους και όποιος θέλει να είναι αυτοπασχολούμενος, με γεια του, με χαρά του, να παραμείνει. Και πολλοί νέοι θέλουν να ξεκινήσουν έτσι. Δεν θέλουμε να απαγορεύσουμε την αυτοπασχόληση. Το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή τα έχει πει κανείς αυτά ε, ε, αυτοπασχόληση θα πρέπει να έχει την ίδια προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα με όλους τους άλλους εργαζομένους. Γιατί αν δεν τους εγγυηθούμε μια στοιχειώδη προστασία, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια ή και αύριο. Αν δεν έχουν ασφάλιση, αν αρρωστήσουν, τι θα γίνει. Αν δεν ασφαλισμένοι απέναντι σε ατυχήματα. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με τους λεγόμενους υποτίθεται αυταπασχολουμένους ε, Uber. Άμα πάθουν αυτοί οι άνθρωποι ένα ατύχημα, τι θα γίνει. Ε, θα πρέπει να σεβαστούμε την αυταπασχόληση, αν είναι γνήσια και ουσιαστική, αν, αν είναι λανθασμένοι, εσφαλμένοι ή ψευδείς, ε, όπου οι άνθρωποι είναι μισοτοί, αλλά τους βαφτίζουν αυτοαπασχολουμένου, θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Madame κυρία Βίντ. Ερώτηση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω δανέζικα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ ε, που ήρθε εδώ και κάθισε εκεί πάνω ψηλά αντί να κάτσει δίπλα μου. Η δική μου ε, ερώτηση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τους εργανόμενους. Ε, η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, απογοητεύτηκε γιατί στην επιστολή της κυρίας Φοντερ Λάιεν, όπου περιγράφει την αποστολή της, δεν ε, μιλάει για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που μας αφορά. Η προηγούμενη Επιτροπή έφτιαξε ένα ε, στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία του 2014-2020 για μηδενικά θανάσιμα ατυχήματα στο χώρο εργασίας. Εσείς ε, θα βρείτε κάποια ευρωπαϊκή, ε, ένα ευρωπαϊκό όραμα για αυτά τα ατυχήματα και για τον καρκίνο που προκαλείται από τον καρκίνο και ε, τι θα κάνετε με το τέταρτο πακέτο των επιβλαβών ουσιών σύμφωνα με την οδηγία για τα καρκινογόνα και τα μεταξυλαξιογόνα. Όταν λέτε ότι θέλετε μια οικονομία που εξυπηρετεί τους ανθρώπους, ε, ένα από τα πρώτα στοιχεία αυτής της οικονομίας είναι να προστατεύει τους εργαζόμενους στην εργασία, τον κόσμο στην εργασία. Είναι σκάνδαλο αυτοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους να εκτίθενται σε κινδύνους ε, για την υγεία τους ή σε ατυχήματα να μην μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, να επιστρέψουν σπίτι τους ε, ασφαλείς γιατί πέθαναν στο χώρο εργασίας. Για μένα λοιπόν η υγεία και η ασφάλεια είναι μια ύψιστη προτεραιότητα. Είπατε ότι δεν είναι στην ε, εντολή μου. Ε, είναι. μιλήσαμε εκεί για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε των πλατφορμών ε, κοιτάξτε, είναι στην αρχή 10 του κοινωνικού πυλώνα. Πρέπει να φτιάξουμε το σχέδιο δράσης, να εφαρμόσουμε τον κοινωνικό πυλώνα. Όταν χρειάζεται πρέπει να υιοθετήσουμε και νομοθετικά μέτρα για να εφαρμόσουμε τον πυλώνα. Άρα συνδέεται άμεσα το ζήτημα αυτό με την υγεία και την ασφάλεια. Δεν μπορεί κανείς ε, να φανταστεί ότι μόλις λήξει το πλαίσιο θα πούμε ότι δεν το χρειαζόμαστε πια. Φυσικά και θα εργαστώ επ' αυτού, θα κάνω προτάσεις στο Κολέγιο των Επιτρόπων και θα επεξεργαστώ νέα ζητήματα που έχουν σημασία για αυτό τον τομέα. Μιλήσατε για τις οδηγίες που σχετίζονται με τον καρκίνο και άλλες ουσίες. Αυτή η συνεργασία έχει ήδη προχωρήσει και πρέπει αυτές τις οδηγίες να τις αναλάβουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε την νομοθετική διαδικασία. Πρέπει να δούμε τις νέες μορφές υγειονομικών κινδύνων, ψυχοκοινωνικών και υπάρχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτή τη στιγμή συζητούμε την ψηφιακή οικονομία. Εκεί, μέσα στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, έχουμε περιλάβει και αυτές τις πτυχές των εργασιακών συνθήκων. Γιατί ε, το θέμα αυτό είναι σημαντικό και η υγεία και η ασφάλεια σχετίζονται και με την ψυχική νόσο που πολλές φορές έχει να κάνει με αυτά. Η επερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Χαίρομαι που άκουσα αυτή την απάντηση από εσά. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας στον χώρο εργασίας, κάθε τέταρτος εργαζόμενος έχει στρες που σχετίζεται με την εργασία του και υπάρχει και ε, κίνδυνος να υπάρχει απώλεια της παραγωγικότητας λόγω των μειοσκελετικών προβλημάτων. Δυστυχώς οι Επιτροπές Μπαρόσο και Γιούνκερ αρνήθηκαν να αναλάβουν δράση σε αυτό το θέμα. Αν εσείς γίνετε επίτροπος, θα προτείνετε νέες πρωτοβουλίες ε, για να βελτιώσετε το εργασιακό περιβάλλον και να προλάβετε το στρες που σχετίζεται με την εργασία. Απάντηση. Μόλις ανέφερα τη νέα οικονομία. Αυτά είναι στοιχεία πτυχές της νέας οικονομίας. Είναι η μετατροπή ε, των εργασιακών συνθήκων ε, στις εταιρείες. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από στρες οδηγούνται και στην αυτοκτονία πολλές φορές. Αυτό το θέμα ε, πρέπει να το αναλάβει η Κομισιόν, αλλά όχι μόνο η Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Οι εργοδότες πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή η κατάσταση είναι βλαβερή όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για την ίδια τους την εταιρεία. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε, πρέπει να βρούμε τις σωστές λύσεις έτσι ώστε το περιβάλλον εργασίας ε, που οδηγεί σε στρες, σε ε, εξάντληση, σε burnout όπως ονομάζεται, σε μειοσκελετικά ζητήματα, ώστε όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολη η λύση. Ως τώρα δεν έχει βρεθεί μια πολύ καλή λύση, όμως το ζήτημα χρειάζει, χρήζει μιας πρακτικής προσέγγισης. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα κουστούμι για όλους. Πρέπει να γνωρίζουμε καταρχάς το θέμα, να συνειδητοποιούμε ότι είναι κακό για όλους, για τον εργαζόμενο, αλλά κυρίως για την εταιρεία. Διότι όταν έχουμε ψυχική νόσο, οι άνθρωποι απέχουν από την εργασία τους όχι για μια μέρα, αλλά για μήνες, για πολύ καιρό. Πρέπει λοιπόν με τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε και είμαι αισιόδοξο ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Η κυρία Μπρουνέ. Μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε και κύριε Σμιτ, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων είναι μια από τις ωραιότερες επιτυχίες της Ευρώπης. Ευνοεί τις ανταλλαγές ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς και δημιουργεί ε, επαγγελματικές ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους, ανήκει νέες αγορές στις επιχειρήσεις και έτσι συμβάλλει στην ευημερία και στην ελευθερία στην Επιρώμα. Ωστόσο, πολλοί ε, Ευρωπαίοι και όλα και περισσότεροι θεωρούν πως δεν επικρατεί δικαιοσύνη και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει εισάγει μια άνηση, έναν άνισο ανάμεσα στο κράτη και ε, ανταγωνισμό στη δικαιοσύνη ανάμεσα στους εργαζόμενους. Δηλαδή, ίδιος μισθός για την ίδια εργασία στην ίδια χώρα μπορεί αυτό να ε, ε, σημαίνει πολύ διαφορετικό κόστος της απασχόλησης. Πώς μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε αυτή την κατάσταση που μπορεί να βλάψει την αίσθηση του ανήκειν στην Ευρώπη. Δύο λεπτά έχετε για την απάντησή σας. Νομίζω πως η ελεύθερη κυκλοφορία ε, υπηρεσιών ε, και παροχών στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντική αρχή όπως είπατε και επιτρέπει ε, τη μετακίνηση όχι για απάτη και κοινωνικό ντάμπινγκ όμως από τη στιγμή όπου υπάρχουν μορφές που κοινωνικού ντάμπινγκ τότε αυτό ε, καθίσταται επιβλαβές. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο με την οδηγία περί αποσπασμένων εργαζόμενων. Το είπα και πριν από λίγο για την αρχή ίδιος μισθός για την ίδια εργασία στο ίδιο ε, μέρος. Τώρα όμως πρέπει σωστά να εφαρμόσουμε και θα έλεγα μάλιστα πολύ πολύ ε, επισταμένα να εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα όχι μόνο για τις χώρες που, που δέχονται ε, εργαζόμενους αλλά και για εκείνες που αποστέλουν, γιατί, ε, που αποστέλουν γιατί δεν μπορεί καμιά χώρα να χρησιμοποιεί κοινωνικό ντάμπινγκ εις βάρος των εργαζομένων της. Αυτό δεν είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πνεύμα και γι' αυτό και υπολογίζω την αρχή εργασίας ε, την επιθεώρηση εργασίας ώστε να εξασφαλίσει πως όλα αυτά τηρούνται και πως οι συνθήκες ανταγωνισμού είναι παρόμοιε, όσο γίνεται πιο κοντινέ. Το θέμα τη κοινωνική πρόνοια είναι περίπλοκο γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε ένα σύστημα όπου έχουμε μία ίδια κοινωνική πρόνοια για όλου. Δεν το επιθυμούμε αυτό. Ο καθένα ε, είναι συνδεδεμένος με το δικό του κοινωνικό σύστημα. Όταν όμως γίνεται παροχή πέρα από τα σύνορα για κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον άνθρωπο αυτό να εγγραφεί στο κοινωνικό σύστημα της άλλης χώρας, γιατί θα έχει δικαιώματα που, τα οποία δεν θα μπορέσει να ε, χαρεί ποτέ. Ε, πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε την κοινωνική ε, πρόνοια σε περίπτωση ελεύθερης ε, παροχής υπηρεσίας. Θα αναλύσουμε την κατάσταση και θα δούμε αν πραγματικά, για, αν γίνεται, λόγω της κοινωνικής ασφάλισης να υπάρχουν να υπάρχουν ε, απαράδεκτες συνθήκες ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Σμιτ. Επί συμπληρωματική ερώτηση, πιστεύετε πως αυτή ε, η κατάσταση κοινωνικής πρόνοιας θα βελτίωνε την κατάσταση όσον αφορά την έλλειψη πολλών δεξιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι η κοινωνική σύγκληση. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη ε, αλληλέγγυα ε, και οικονομική ανάπτυξη ε, μόνο, αλλά και για την κοινωνική ανάπτυξη, γιατί η υπόσχεση της Ευρώπης είναι τελικά κοινή ευημερία για όλους. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε ο καθένα εκεί όπου κατοικεί θα μπορεί να έχει συνθήκε εργασία ε, σωστέ. Όμω ταυτόχρονα ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την ελεύθερη κυκλοφορία. Είδαμε λοιπόν ότι σήμερα υπάρχουν 17 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που ζουν σε διαφορετική χώρα από τη χώρα προέλευση του και ζώντα συχνά σε μια άλλη χώρα έχουν και εργαστεί σε αυτή και βοηθούν ε, στην καταπολέμηση της έλλειψης εργατικού δυναμικού που μπορεί να υπάρχει εκεί στη χώρα υποδοχή. Αυτό είναι προ όφελο όλων. Αλλά η ελεύθερη κυκλοφορία δεν μπορεί να σημαίνει αναγκαστική ελεύθερη κυκλοφορία. Θα πρέπει να είναι θελοντική. Μια ελεύθερη κυκλοφορία η οποία θα ωφελεί τόσο τον άνθρωπο τον ίδιο όσο το χώρα ε, ε, υποδοχής όσο και τη χώρα ε, αποστολής. Μόνο έτσι θα έχουμε αλληλεγγύη. Ο κύριο Φέρμπερ, συνάδελφο από την Οικονομική και Νομισματική. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να μιλήσω γερμανικά. Αξιότιμη κύριε Σμιτ, ε, στην επιστολή ε, αποστολή σα, ε, γίνεται λόγο για μια αντασφάλιση του επιδόματο ανεργία στην εισαγωγή σας μιλήσατε έτσι γενικώ για μακροοικονομικούς σταθεροποιητές. Πώς φαντάζεστε μια τέτοια αντασφάλιση των επιδομάτων ανεργία, για να αποφευχθεί αυτό που ονομάζουμε ηθικό κίνδυνο, moral hazard. Δηλαδή να κάνουμε έτσι γενικά και αόριστα υποσχέσεις και τελικά να μην χρειάζεται να λογοδοτούμε για αυτές. Πώς το φαντάζεστε όλο αυτό το σύστημα. Απάντηση στα γερμανικά. Καταρχάς θα έλεγα ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις προϋποθέσεις. Πότε θα ε, τίθεται σε ισχύ, κινητοποιείται στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η αντασφάλιση. Αυτό θα πρέπει να το ορίσουμε. Ποιο θα είναι εκείνο το οικονομικό σοκ, ο κραδασμός που θα πούμε ότι τώρα κινητοποιείται αυτός ο μηχανισμός αντασφάλισης των επιδομάτων ανεργίας. Αυτές είναι παράμετροι που θα πρέπει από κοινού να ορίσουμε. Και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην έχει υπάρξει στο παρελθόν ο ηθικός κίνδυνος. Αυτό είναι το ερώτημα και το ζήτημα. Δεν είναι ότι αυτό το μέσο θα προκαλέσει ηθικό κίνδυνο. Ε, θα συνεισέφερε μάλλον να ενισχυθεί ο προηγούμενος προϋπάρχον ηθικός κίνδυνος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να κάνουμε μια καλή δημοσιονομική πολιτική και ξέρω ότι εσείς αγωνίζεστε πολύ σχηρά γι' αυτό και να υπάρχουν και κανόνες που να σέβονται τα κράτη-μέλη, είναι υποχρεωμένα, είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ψηφεί τους κανόνες και μετά να υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο να επικαλείται για να σωθεί. Δεν είναι καθόλου ε, το νόημα και ο σκοπός. Αλλά υπάρχουν κραδασμοί στην οικονομία μας που μπορεί να υπάρξουν και να είναι και ασύμετροι πολύ συχνά. Ε, τι να κάνουμε. Αυτό δυστυχώς είναι στοιχείο και συστατικό του οικονομικού μας συστήματος και θα πρέπει εμείς αυτούς τους κραδασμούς να τους απορροφούμε κάπως και όχι να έχουμε μόνιμες μεταβιβάσεις πόρων από τους μεν στους δε, αλλά να εξασφαλίζουμε όταν υπάρξει ένας τέτοιος κραδασμός να μην βυθιστεί ε, σε ένα απίθμανο χάος η οικονομία Τη χώρας αυτή και οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια κοινωνική εξασφάλιση ακόμα και αν αντιμετωπίζει μεγάλε δυσκολίε το κράτο του για να το κάνει αυτό για λόγου δημοσιονομικού και χρηματοοικονομικούς και αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο συγκεκριμένο μέσο. και είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε κύριε Φέρμπερ πολύ συγκεκριμένα αν κοιτάξετε την οικονομική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία στα κράτη-μέλη, Πού συγκεκριμένα θα λέγατε ότι να μια περίπτωση που θα μπορούσε να έχει κινητοποιηθεί αυτή η αντασφάλιση των επιδομάτων ανεργία. Σε ποια συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω συγκεκριμένε περιπτώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ δίκαιο να αναφερθώ σε παραδείγματα και να κατονομάσω. Κοιτάζοντα πάντω την τελευταία κρίση, ε, σε διάφορες χώρες το πρόβλημα δεν ήταν ότι είχαν τεράστια ελλείμματα δημοσιονομικά παράγει, αλλά ήταν θύματα της κρίσης παρόλο που στην αρχή ήταν πάρα πολύ ε, σταθερές οικονομίες και είχαν μάλιστα και πλεονάσματα και ξέρετε και ποια χώρα έχω στο μυαλό μου και ε, είναι και νότιες χώρες αυτές οι οποίες επλήγησαν σφοδρότατα από την κρίση αυτή και τα πρώτα θύματα ήταν οι νέοι, οι νέοι οι οποίοι δεν βρήκανε δουλειά. Ε, ε χάσαν τη δουλειά τους και ήταν τα πρώτα θύματα. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την εγγύηση για την νεολαία. Παρακαλώ. Ε, κύριε Φέρμπερ, τώρα τι θα γίνει. Ε, δεν έχουμε και επερώτηση της επερώτησης, σχόλια και παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή. Η κυρία Νίνα Γκίν και πάλι από την Οικονομική και Νομισματική για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε Σμιτ, ε, Διαγράψατε το ρόλο της κοινωνικής οικονομίας στην αντιμετώπιση της ανέχειας και τη μείωση των ανισοτήτων. Χαιρετίζω τη μεγαλύτερη έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινωνική οικονομία, γιατί θεωρώ ότι αυτή ε, τρέφει εναλλακτικά συστήματα. Ένας από τους βασικούς, μια από τις βασικές ανησυχίες μας. Ε, ποια θα ε, είναι ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας ε, και μέσα στη βιώσιμη μετάβαση. Πώς θα συνδυάσετε τις επενδύσεις με τις κοινωνικές κοινωνικές ανάγκες. Και θέλω και να συνεχίσω από αυτό που είπε ο Μάρκους Φέμπερ σχετικά με το ε, ε, πρόγραμμα αντασφάλισης. Ε, πώς θα μαζέψετε την υποστήριξη των κρατών μελών πως τώρα αντιτίθεντο αυτό και πώς θα διασφαλίσετε ότι αυτή η αντικυκλική λειτουργία σταθεροποίησης θα υποστηρίξει τα εθνικά συστήματα ανεργίας όταν υπόκεινται σε στρες και θα τα δίνει κίνητρα να ενισχυθούν χωρίς να τιμωρούνται ε, με όρους τα κράτη-μέλη. Το πρώτο που αναφέρατε για την κοινωνική οικονομία. Σε όλη την Ευρώπη ήδη έχουμε μια πολύ ενεργή κοινωνική οικονομία που δρά στις περιφέρειες, ε, στις περιοχές, στην επικράτεια όπου ε, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς που τις χρειάζονται περισσότερο. Έχουμε ε, φροντίδα για τα παιδιά, φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Αυτό είναι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας μας, ένας τομέας που πρέπει να ενισχύσουμε. Όχι μόνο γιατί παρέχουμε ε, υπηρεσίες κοινωνικές, αλλά γιατί δημιουργούνται ενεργά και θέσεις εργασίας. Στην κρίση είδαμε ότι σε αυτόν τον τομέα δεν καταστράφηκε καμία θέση εργασίας. Μάλιστα δημιουργήθηκαν νέες θέσεις χωρίς ένα ε, πρόγραμμα αντασφάλισης της ε, ανεργίας. Οι επενδύσεις είναι σημαντικές σε αυτό το τομέα. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να, να γράψει ε, και να μιλήσει στο πρόγραμμα Juncker, να δώσει δάνεια στην κοινωνική οικονομία. Αυτό είναι μια σημαντική αναγνώριση του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ στις κοινωνικές επενδύσεις. Αν θέλουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, θέλουμε και σταθερές κοινωνικές συνθήκες, που σημαίνει κοινωνική επένδυση στην εκπαίδευση, στη φροντίδα των παιδιών και στην υγεία. Αυτό συνιστά μια ε, καλή οικονομία όταν έχει ένα σταθερό κοινωνικό περιβάλλον. Επενδύσεις λοιπόν στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι σημαντικές. Και στη νέα οικονομία υπάρχει ε, μια διασύνδεση με αυτό και με τη νέα οικονομία, διότι υπάρχει το τομέας της αεφορίας όπου είναι ιδιαίτερα ενεργή η νέα οικονομία, τα νέα μοντέλα της ενέργειας για παράδειγμα, για το πρόγραμμα της ανεργίας. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να πείσουμε και να αφαιρέσουμε τις κατανοητές ε, ε, ανησυχίες ε, που έχουν κάποιοι. Δεν θέλουμε να ενισχύσουμε τον ηθικό κίνδυνο, γιατί πραγματικά είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των χωρών που ωφελούνται, αλλά και όλων των χωρών, ειδικά ε, όταν υπάρχει μια ε, σταθερή οικονομική και νομισματική ένωση. Επερώτηση. Ναι, για το θέμα της ανεργίας αναφερθήκατε στις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και της τεχνικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας. Το 50% των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη είτε θα αλλάξουν είτε θα εξαφανιστούν. Υπάρχουν άνθρωποι με λίγες δεξιότητες. Ποια μέτρα εσείς θα θεσπίσετε ως επίτροπος για να αντιμετωπίσετε αυτό το χάσμα δεξιοτήτων που υφίσταται ήδη. Και λαμβάνοντας υπόψη ε, και το γεγονός ότι χρειάζεται μια ισότητα, ε, ειδικά στον τομέα του εμπορίου. απάντηση. Δεν θα συζητήσω το 50% αλλά σίγουρα οι επιπτώσεις της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής μεταμόρφωσης, οι επιπτώσεις της θα είναι σοβαρές, βαριές. Θα υπάρχουν όμως νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν και αυτές ο κόσμος θα μπορέσει να τις πάρει μόνο όταν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. Η ε, επιμόρφωση, οι νέες δεξιότητες, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων είναι σημαντικά στοιχεία του μέλλοντος. Θα πρέπει να έχουμε τη σωστή εκπαίδευση, να έχουμε αναβάθμιση των δεξιοτήτων, να αλλάξουμε τις δεξιότητές μας έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε αυτές που εξαφανίζονται για να μπορέσουμε να αναλάβουμε τις νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε περισσότερο στο upskilling και στο reskilling. Πρέπει το ESF Plus να δώσει περισσότερα χρήματα για αυτόν τον κλάδο. Είναι θέμα κεντρικής σημασίας και πρέπει να ενσωματωθεί και, και στις ε, συστάσεις αναχώρα. Κάτι που έχει ήδη γίνει στο εγγύς παρελθόν. Η επένδυση περισσότερων χρημάτων στο στους ανθρώπους. Έχουμε την ατζέντα για τις δεξιότητες ε, η νέα πρόεδρος της Κομισιόν. Ε, μου έχει ζητήσει να αναθεωρήσω, να αναδιαμορφώσω αυτή την ατζέντα. Ευχαριστούμε που απαντήσατε την επερώτηση που τελικά δεν ήταν επερώτηση, ήταν ερώτηση. Θα ζητήσω ευγενικά από όλους εσάς ε, να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας σε σχέση με το χρόνο. Έχουμε αργήσει πολύ σε αυτό το στάδιο, παρακαλώ. Η απάντηση και η ερώτηση είναι ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Λιγότερα σχόλια, περισσότερες ερωτήσεις παρακαλώ. Επόμενος ο κύριος ε, Σατούρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συμφωνούμε όλοι εδώ ότι η ευρωπαϊκή υπόσχεση θα πρέπει να βασίζεται σε δύο βάθρα. Ε, δουλειά για όλους και προστασία για όλους. Ε, οι οικονομικοί παράγοντες ε, τα κανονίζουν για να ε, ραπετεύουν και από τα δύο. Βαφτίζουν τους μισθωτούς αυτοπασχολούμενους, έχουν μια σχέση εργασίας χωρίς να σέβονται τα δικαιώματα, το εργατικό δίκαιο με επισφάλεια, δεν σέβονται τίποτα, ούτε ωράρια, ούτε ασφάλεια και ταυτόχρονα με διάφορες υπεργολαβίες ε, κανονίζουν να μην είναι κανένας υπεύθυνο. Όταν έχουμε ατυχήματα και όταν έχουμε κρίσεις, είναι τέτοια η αλυσίδα των υπεργολάβων, όπου δεν γίνεται σεβαστό αυτό το βάθρο το κοινωνικό. Θέλω να μου απαντήσετε συγκεκριμένα, κύριε υποψήφια Επίτροπε, για αυτά τα δύο. Θα φέρετε νομοθεσία για να ενισχυθεί ε, η εφαρμογή του εργατικού δικαίου παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχυθεί και η ευθύνη και η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, ό,τι τεχνάσματα και να βρίσκουν με αλυσίδες υπεργολάβων, ε, για να μην όταν υπάρχει μια δυσκολία να ξέρουμε ποιο είναι ο πρώτος ε, που έχει δώσει την εντολή και να τον φέρουμε απέναντι στι ευθύνε του και να εφαρμοστεί το δίκαιο. Πολύ συγκεκριμένα για την πρώτη ερώτηση, ε, για τους υπεργολάβους. Η πρώτη οδηγία που τροποποιεί την απόσπαση ορίζει ρητά την ευθύνη των υπεργολάβων και εκείνων που τους κάνουν την ανάθεση. Είναι η αλυσίδα, πολύ ωραία την περιγράψατε, οι ευθύνε θα πρέπει να εντοπίζονται ξεκάθαρα. Και εκεί περιμένω από την Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης ε, να παρακολουθεί αυτές ε, τις περίεργες κατασκευές και τις σκοτεινές ε, για να διαχέεται η ευθύνη και να εξαφανίζεται των διαφόρων εις βάρος των εργαζομένων που αποσπώνται από χώρες με εικονικές εταιρείες, ταχυδρομικές θηρίδες και πάει λέγοντας. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε αυτό, να το αναπτύξουμε, αλλά εκεί χρειάζεται να εφαρμόζονται στο ακέραιο κανόνες που ήδη υπάρχουν για την καλή εργασία ποιοτικά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ιδέα του ανταγωνισμού όλοι εναντίον όλων δεν μπορεί να είναι τα θεμέλια του οικονομικού μας συστήματος, ούτε είναι. Και εκεί πιστεύω ότι το συνειδητοποιούμε σιγά σιγά αυτό. Και θέλουμε να ξαναβρούμε τις αρετές ε, αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε πραγματική γνήσια οικονομία, κοινωνική οικονομία της αγοράς, με δικαιώματα και με κοινωνικές διαπραγματεύσεις συλλογικέ με κοινωνικά δικαιώματα για κάθε κατηγορία εργαζομένων, μισθωτών. Μιλήσαμε για τις πλατφόρμες, μιλήσαμε για την απόσπαση των μισθωτών, που δεν μπορούν να είναι ε, όμοιροι οποιασδήποτε κατάστασης και να υπάρχει έλεγχος. Βεβαίως υπάρχουν κατακρίσεις, αλλά κάθε φορά θα πρέπει να αναρωτιόμαστε πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα περιορίσουμε ε, και πώς θα καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτές τις καταχρήσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν νέες μορφές εργασίας, αυτοπασχολούμενοι πολύ συχνά αναγκαστικά, που δεν, δεν ξέρουν καν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μισθωτοί και είναι αυτοπασχολούμενοι, με διάφορες εξωτερικές αναθέσεις εργολαβικούς εργαζόμενους κτλ. Εκεί θα εστιάσουμε την επόμενη πενταετία. Επερώτηση, ευχαριστώ. Ε, έχω την αίσθηση, αλλιώς διορθώστε με, ότι όταν υπάρχει εξωτερική ανάθεση και υπεργολαβία, ο έλεγχο εφαρμογή των κανόνων είναι εθνική αρμοδιότητα. Αν θέλουμε να υπάρξει ευρωπαϊκή αρχή, δεν μπορούμε να επαφιέμεθα στα κράτη-μέλη να κάνουν του ελέγχου. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε προς μια ευρωπαϊκή αρχή που να κάνει τους ελέγχου και την επιθεώρηση σε επίπεδο κεντρικό. Νομίζω ότι η Ευρώπη γίνεται πάντα σταδιακά και βήμα-βήμα η οικοδόμηση της Ευρώπης δηλαδή. Ε, τώρα δημιουργείται μια αρχή απασχόλησης. Ε, θα πρέπει ε, πρώτα απ' όλα να ε, μας δώσει ένα σημαντικό εργαλείο. Γιατί η αρχή για την απασχόληση συγκεντρώνει τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία και του Κοινοβουλίου, αλλά κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή λοιπόν μπορεί να οργανώσει επιθεωρήσεις επιτόπου, ακριβώς όπου μπορεί να εμφανίζονται τέτοιες πρακτικές και μετά να κάνει προτάσεις για να ε, καταπολεμούμε αποτελεσματικά αυτές τις καταχρήσεις και τις εκτροπές. Τα κράτη επίσης θα πρέπει να έχουν μέσα και πόρους. Διαπιστώνω ότι οι πάντες διαμαρτύρονται για το κοινωνικό ντάμπινγκ και μιλώ και για τη χώρα που γνωρίζω ακόμα αρκετά καλά, οι πόροι και οι ανθρώπινοι και οι οικονομικοί των επιθερήσεων εργασίας δεν έχουν αυξηθεί, για να μην πω ότι μειώθηκαν κιόλας. Αυτά συμβαδίζουν. Δεν μπορούμε από τη μια να καταγγέλουμε τον κοινωνικό ντάμπινγκ και να μην έχουμε τα μέσα να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, να παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά επί τόπου τελικά να πιέζει τα κράτη-μέλη για να ελέγχουν, να συνεργαζόμαστε στις επιθεωρήσεις. Τώρα το να παίξει η Ευρώπη αυτό το ρόλο, να τον αναλάβει. Κάντε λίγη υπομονή, όχι ακόμα. Ε, κυρία ε, Ρίση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Κύριε Σμιτ, με την παρέμβασή μου θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα-δύο θέματα που σχετίζονται με τα σύνορα και η διασυνοριακή εργασία σύμφωνα με το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και η μετατόπιση ε, μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, είναι γνωστό ότι το περασμένο Μάρτιο το κείμενο δεν έτυχε της ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο λόγω της ε, ε, αντίθεση ορισμένων χωρών όπως το Λουξεμβούργο μεταξύ αυτών. Πώς σκοπεύετε να συνδυάσετε την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας σας με την ε, ε, πολιτική ε, την ομοιόμορφη που προτείνει και προωθεί η Κομισιόν ε, για τα κοινωνικά θέματα. Τώρα, το θέμα της μετατόπισης και της κινητικότητας των εργαζόμενων και της απόσπασης των εργαζομένων μέσα στα ίδια τα κράτη μπορούν να αποτελέσουν μορφή κοινωνικού ντάμικα ανάμεσα στα κράτη και εντός των κρατών. Σκοπεύετε να ευνοήσετε νέες βιομηχανικές πολιτικές που να προλαμβάνουν τη μετατόπιση και το κοινωνικό ντάμπινγκ. για την πρώτη ερώτηση. Όντως δεν υπήρξε ε, ειδική πλειοψηφία. Αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω πως δεν είναι το Λουξεμβούργο το οποίο έκανε, το, δημιούργησε το πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε και τόσο πολύ βάρος αλλά εγώ είμαι υποψήφιος επίτροπος, δεν είμαι Έλληνας Λουξεμβούργιος που μάλιστα έχει φιλοδοξία να γίνει Ευρωπαίος. Ε, ε, ε, είμαι ένας Λουξεμβούργιος που θέλει να γίνει Ευρωπαίος επίτροπος και αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κοινό συμφέρον, το ευρωπαϊκό συμφέρον. Χάρη λοιπόν στο Στην επιμονή της Κομισιόν θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση για το 883, να εξασφαλίσουμε ίση και προστασία και δυνατότητα μετακίνησης των εργαζομένων ώστε να μην παρεμποδίζονται από τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης. Τώρα, επίσης έχουμε εισάγει μια ολόκληρη σειρά μέτρων. Ε, έχουμε μιλήσει για την οδηγία, για την απόσπαση. Τώρα θέλουμε να εξασφαλίσουμε και τη σωστή εφαρμογή ε, αυτής της οδηγίας. Δηλαδή δεν θέλουμε να δημιουργούμε κάθε φορά ένα νέο νομικό μέσο ή νομοθετικό μέσο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εφαρμόζεται σωστά, ε, με μεγάλη επιμέλεια. Ε, το νομοθέτημα που έχουμε ήδη εγκρίνει, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε νέες μορφές κοινωνικού ντάμπινγκ, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε σύντομα, ώστε, γρήγορα, ώστε να αντιδράσουμε σε αυτές τις νέες μορφές κοινωνικού ε, dumping. Πάντως τώρα έχουμε ένα καλό, πολύ καλό εργαλείο, θα πρέπει σωστά να εφαρμαστεί, επαναλαμβάνω, και η αρχή της εργασίας είναι ένα νέο μέσο που έχουμε στη διαθεσή μας, πρέπει να το κάνουμε να ενεργήσει αποτελεσματικά. Περώτηση. κοινωνικό ντάμπινγκ και ε, αθέμητος ανταγωνισμός που γίνεται ανάμεσα ε, στις χώρες, ας πούμε στην Ιταλία και τις ε, όμορες χώρες. Για να περιορίσουμε τον αγώνα μείωσης προς τα κάτω των μέτρων προστασίας και των αποφάσεων που λαμβάνονται μέσω των διάφορων project, ας πούμε το πολιτικό project της Ursula von der Leyen, μπορείτε να μας διευκρινίσετε πώς σκοπεύετε να προσαρμόσετε τις μισθολογικές πολιτικές μέσα στα κάτι μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ε, υπάρχουν μεγάλες ε, ε, ανισορροπίες στο κόστος εργασία που ακριβώς βρίσκονται και στη ρίζα της μετατόπισης των εργαζόμενων, αλλά και στη ρίζα μεγάλων ανισοτήτων όσον αφορά την απασχόληση και την αγορά. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. Πιστεύω πως ήδη υποδείξατε τι πρέπει να γίνει, διότι φιλοδοξία μας είναι να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε την κοινωνική σύγκληση. γιατί ακόμα και μια Ευρώπη δυναμική και ανταγωνιστική δεν μπορεί να επιδίδεται σε ξέφρενο ανταγωνισμό για το ποιος θα έχει τους χαμηλότερους μισθούς. Νομίζω πως αυτό ε, θα υπάρχει πάντοτε ε, κάποιες περιοχές δηλαδή όπου στον κόσμο που η μισθή θα είναι χαμηλότερη. Όταν μιλάμε για ένα πλαίσιο για το μίνιμουμ ε, εισόδημα που θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια κάποια σύγκληση μισθολογική στην Ευρώπη, Σύγκληση δεν σημαίνει ταυτότητα. Σύγκληση δεν σημαίνει μήνυμο με μισθώσεις στη Βουλγαρία να έχουμε ίδιο μισθό στη Γαλλία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και στη Γερμανία. Αλλά ε, σημαίνει προσέγγιση η σύγκληση. Να έχουμε κάπως ε, ε, σχετικούς μισθούς. έχει αυτό αντίκτυπο σε όλους τους μισθούς και θα επιτρέψει να καταπολεμήσουμε και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Κυρία Σιλδε, εσείς τώρα. Ευχαριστώ μεταξύ των ευθυνών που και των αρμοδιοτήτων που θα αναλάβετε είναι η εγγύηση για το παιδί. Η δική μας προτεραιότητα πρέπει να είναι να πατάξουμε την φτώχεια, την ανέχεια και χάρη στα μέτρα που εμείς λάβαμε στην Πολωνία καταφέραμε να μειώσουμε την ανέχεια κατά 50%. Εσείς στις απαντήσεις σας είπατε ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση των παιδιών θα πρέπει φυσικά να βελτιώσουμε και την κατάσταση των οικογενειών. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν αυτό καλύπτει και να, πάρεις, να παίρνεις παιδιά από τους γονείς τους, όπως κάνει το Jungentamt, να παίρνουν τα παιδιά δηλαδή από την οικογένειά τους ε, χωρίς κάποια αιτιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν όμως αρνήθηκε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τι θα κάνετε με αυτό το πρόβλημα. La γιατί αρνήθηκε η Επιτροπή, είναι απλό γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ δεν μπορώ να αποφανθώ για την τάδε ή τη δίνα υπόθεση. Φυσικά υπάρχουν υποθέσεις όπου το συμφέρον του παιδιού είναι να μην μείνει με τους γονείς. Αυτά είναι ειδικέ ε, περιπτώσεις και δεν θα ορίσει ε, δεν θα ορίσουν οι Βρυξέλλες ποιος ε, και πότε θα έχει το παιδί και υπό ποιους όρους. Νομίζω ότι αυτό εναπόκειται ξεκάθαρα στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και των υπηρεσιών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Τώρα για την εγγύηση για το παιδιά θα αναλάβουμε κάθε είδους δράση που θα ενισχύει την ισότητα ευκαιριών για τα παιδιά, την επένδυση στα παιδιά. Όλα αυτά ε, τα χαιρετίζουμε και όλα αυτά θα τα επιδείξουμε σε αυτούς που θα είχαν συμφέρον να ακολουθήσουν ένα τέτοιο παράδειγμα. Κυρία Σιλόφ, έχετε επερώτηση. Μιλάμε για τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, οπότε δεν θεωρείτε ότι αυτή η συνεργασία με τα κρήτα κρατών μελών θα ήταν απαραίτητη μια τέτοια συνεργασία. Γιατί οι Ευρωπαίοι που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για βοήθεια είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντιμετωπιστεί ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν θεωρείτε λοιπόν ότι η Επιτροπή όπως και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρουν στα χέρια τους αυτό το θέμα και να κάνει κάτι η Κομισιόν σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Επαναλαμβάνω όλη μια φορά. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Δεν είναι η αρμοδιότητα της Κομισιόν να επέμβει άμεσα. Τώρα, αν υπάρχουν υποθέσεις μεταξύ κρατών μελών ε, που είναι αντίδικοι ή τέλος πάντων έχει να κάνει με το εφαρμοστέο οικογενειακό δίκαιο σε πολλά κράτη-μέλη, ίσως μπορούμε να εξετάσουμε πώς θα μπορούσαμε να επιλύσουμε μια κατάσταση που προκύπτει, γιατί ε, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε υπάρχουν πολλές οικογένειες ε, που οι γονείς είναι από διαφορετική χώρα και εθνικότητα. Έτσι λοιπόν το οικογενειακό δίκαιο των μεν ή των δε πρέπει να εφαρμόζεται σωστά υπέρ, υπέρ του συμφέροντος του παιδιού πάντα. Υπάρχει σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτή πρέπει πάντοτε να γίνεται σεβαστή, να την τηρούμε. κύριος παρακαλώ. Αγαπητέ Επίτροπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για την ανεξάρτητη διαβίωση κάνει hearing, ακρόαση αυτή την εβδομάδα. Ε, δεν χρειάζεται να πω την επίκαιρη ερώτησή μου. Θα ήθελα να μάθω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προβλέπει ε, μέτρα για την στρατηγική για ανθρώπους με αναπηρία 2020-2030 ε, ε, μέτρα ε, που προωθούν την συμπερίληψη, την κοινωνική ένταξη και τις κοινωνικές επιχειρήσεις για μεταφορές προσβάσιμες από και προς το χώρο εργασίας, την ανάπτυξη, την κατάρτιση και φυσικά ε, και προφανώς προσβάσιμους χώρους εργασίας. Ε, I think we Πιστεύω ότι πρόσφατα έχουμε εγκρίνει ε, την πράξη για την προσβασιμότητα που είναι πρόοδος και βοηθάει και τα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό τους βίο. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι, πολιτικές, οι πολιτικές μας για την απασχόληση θα πρέπει να εστιάζουν περισσότερο σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και αν κοιτάξουμε τα αριθμητικά στοιχεία θα διαπιστώσουμε πραγματικά ότι άνθρωποι με αναπηρίες είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες ή μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον εργασιακό τους χώρο και στην αγορά εργασίας. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες και γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες, διότι τα εκπαιδευτικά μας συστήματα ήδη δεν ε, ευνοούν ε, τους ανθρώπους με αναπηρία. Δεν έχουν καν τις ευκαιρίες να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες από τα εκπαιδευτικά μας συστήματα που δεν ε, είναι προσαρμοσμένα με τις δικές τους ανάγκες. Και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξει διάκριση γιατί είναι από τις βασικές μας αρχές η έλλειψη διακρίσεων. Και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ακριβώς τις ίδιες ευκαιρίες ε, στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους και μέσα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στις πολιτικές που συμπεριλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες των ε, πολιτών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ε, στον εργασιακό χώρο και στην αγορά εργασίας. Και μεταξύ αυτών είναι και τα άτομα με αναπηρίες. Είναι πραγματικός στόχος αυτός για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμού στην οποία ε, φιλοδοξούμε. και θέλω να είναι και σημαντικός ε, στόχος και σκοπός των επόμενων ετών αυτός. Να δίνουμε την ευκαιρία σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων με αναπηρίες. Και πρέπει να πω ότι οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν εκεί. Είναι ο σωστός τρόπος αυτός. Θα πρέπει όμως να υποστηρίζουμε τους ανθρώπους για να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τις ψηφιακές. Και είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε τουλάχιστον να μειώσουμε ε, σε μεγάλο βαθμό τα ελλείμματα. Συμπληρωματική ερώτηση. Πιστεύετε ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη θα μπορούσε να είναι κατάλληλο εργαλείο για να δώσει κίνητρα στους εργοδότες να ε, απασχολούν ε, εργαζομένους με αναπηρίες. Προβλέπετε μέτρα για τους εργοδότες να μπουν ε, σε αυτό το δρόμο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις σας. I'm I'm a believer. Εγώ πιστεύω στην κοινωνική εταιρική ευθύνη αλλά ταυτόχρονα δεν περιμένω και τα πάντα από αυτήν. Θα πρέπει και εκεί να υπάρχουν κάποιοι κανόνες και να υποχρεούνται οι εργοδότες να σέβονται τους κανόνες αυτές. Υπάρχουν χώρες που έχουν και ποσόστοση. Δεν ξέρω, 5% δεν θυμάμαι πόσο στο Λουξεμβούργο. Ε, υπάρχει ποσόστοση για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία. Ε, θα πρέπει όμως να έχουμε ένα ε, όραμα για μια κοινωνία με μεγαλύτερη συνοχή, για να έχουν όλοι καλές ευκαιρίες. Και έχω δει σε πολλές περιπτώσεις, όταν ήμουν ακόμα υπουργό Εργασίας, ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στις ικανότητες που έχει ε, κάποιος με αναπηρία. Μπορεί να είναι εξίσου ικανή να μην πω και παραγωγικότεροι πολλές φορές γιατί έχουν περισσότερα κίνητρα. Βεβαίω, να εθαρρύνουμε τι επιχειρήσει και του επιχειρηματίε, να τους πιέσουμε λίγο και να του βοηθήσουμε κιόλα, γιατί ε, ε, χρειάζονται προσαρμογέ ε, στο χώρο εργασίας. Φυσικά θα πρέπει όλα αυτά να τα προωθήσουμε. Oh, thank Κύριε Αλσαλάνη, θα μιλήσω σου ειδικά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ καταρχά Επίτροπε για τις ε, γραπτές και τις προφορικές σα απαντήσεις. Ε, ε, συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας για αυτά τα θέματα. Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σέβεται την ισότητα των κρατών μελών, καθώς και την εθνική τους ταυτότητα που εκφράζεται στα συντάγματά του. Η αρμοδιότητες λοιπόν περιορίζονται από την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Ακριβώς για τα θέματα της απασχόλησης έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση στην Σκανδιναβία. Είπατε ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε, να διορθώσουμε αυτό που δεν είναι χαλασμένο. Όμως όταν βλέπει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εντύπωση πως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή συντονισμός δεν σημαίνει εναρμόνιση. Πώς θέλετε συγκεκριμένα λοιπόν να εγγυηθείτε το σεβασμό των εθνικών διαφορών και την αυτονομία των εταίρων μέσα στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων. Well, I can only repeat what I've said. You know... Δεν μπορώ παρά να παραλάβω τα όσα είπα. Εγώ είμαι ο οπαδός της υπηκουρικότητας και είμαι ο παδόν και μπορώ να το πω των κοινωνικών συστημάτων που βασίζονται σε τον ισχυρό κοινωνικό διάλογο και τους ισχυρούς κοινωνικούς εταίρους και θα ήταν πραγματικά παράλογο να παρέμβει κανείς σε αυτά τα συστήματα ή να προσπαθήσει να τα αλλάξει. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν προτείνουμε ένα πλαίσιο για μήνυμο μισθούς, θα υπάρχουν και οι εγγυήσει εκεί που, για όλα τα συστήματα που βασίζονται στι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω, μπορώ να σα πω αυτή την εγγύηση και να είστε βέβαιοι ότι θα μιλήσουμε με του συναδέλφου και στην Κομισιόν που επίση άμεσα ε, ασχολούνται με αυτά τα θέματα και που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι, αλλά και θα συζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με όσους εδώ είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα ζητήματα. Ε, αρκετοί από εσά ήδη το αναφέρατε και μετά θα πάμε σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένες της Σουηδίας αλλά και των υπολείπων χωρών ώστε να συζητήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα μπορέσετε να διατηρήσετε το σύστημα το οποίο σας είναι τόσο προσφυλές. Σας ευχαριστώ για αυτήν σας την απάντηση. Όντως, ε, πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε εδώ ε, ευχαριστημένοι, αλλά ε, θα πρέπει να κατανοήσετε πως αυτό το μοντέλο για μας είναι εξαιρετικά ριζωμένο γιατί βασίζεται στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας και διαπιστώνουμε πως επικρατεί μία νομική κατάσταση η οποία είναι εδρεωμένη, παγιωμένη στη χώρα μας. Πώς θέλετε λοιπόν να ενθαρρύνετε και στις υπόλοιπες χώρες τον κοινωνικό διάλογο. Κατά τα λοιπά, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Έχετε ένα λεπτό για απάντηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, μάλιστα. Εγώ νομίζω πως όταν μιλάμε για πλαίσιο, για νομικό πλαίσιο, για τα ελάχιστα ημερομίσθια, δεν θα γινω, μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο να γίνει χωρίς να μιλήσουμε με τους κοινωνικούς εταίρους. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά πρέπει να στραφούμε και στους κοινωνικούς εταίρους μεμονωμένα στα κάτι μέλη. Ιδιαίτερα εκείνος που είναι τόσο ευαίσθητη για αυτά τα θέματα και λόγους που εσείς αναπτύξατε. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις μας θα διατηρούν το σύστημα. Διότι δεν είναι θέμα το να, μετα... το να μετατρέψουμε, να αλλάξουμε το σύστημα. Αλλά στόχος είναι να σας διαβεβαιώσω και να σας καθησυχάσω πως δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση και ούτε θα αποκτήσω τέτοια πρόθεση. Λοιπόν. Κύριε Πάντων, η ερώτησή σας. Συμφωνεί ο Επίτροπος με μένα ότι στο θέμα των ε, ε θέσεων εργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεσμικά ρατσιστική παρά τις σα ε, ότι θα έχετε αξιοπρεπή ε, ε, θέση εργασία για, εργασίας για όλους δεν έχετε κάποιο σχέδιο για τις εθνοτικές ε, μειονότητες, ε, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ε, υπόκεινται σε διακρίσεις στο χώρο εργασίας. 76% των ανθρώπων που δεν είναι σε κατάρτιση, εκπαίδευση ή εργασία είναι από αυτές τις κατηγορίες. Εδώ στο Βέλγιο το 1 τρίτο των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί στο Βέλγιο είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε σχέση με τεράστια ποσοστά αφρο, αφροαμερικανικών ανθρώπων από τις αφρικανικές χώρες που δεν έχουν τέτοια εκπαίδευση. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην διαφορετικότητα, αλλά αυτό γίνεται μόνο όταν κανείς είναι άσπρος. Είχαμε την Western και μια οργάνωση, μια ε, ε, ένα θεσμό της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα κράτη-μέλη λοιπόν να ακούν τον Επίτροπο ή την Επιτροπή όταν στο σπίτι τους, στα του οίκου τους, δεν είναι σωστή. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θεσμικά ρατσιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο λεπτά για την απάντηση. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι η έλλειψη διακρίσεων αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δεν είμαι αφελής. Δεν είμαι καθόλου αφελής. Ξέρω ότι υπάρχουν ευάλωτοι πληθυσμοί που υποφέρουν και στην αγορά εργασίας. Και πραγματικά, δεν έχουμε μόνο καλές αρχές. Πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα για να εφαρμόσουμε αυτές τις καλές αρχές παντού συμπεριλαμβανομένων των δικών μας επιχειρήσεων, των θεσμών μας, οπουδήποτε. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει επίσης την Ευρώπη και πρέπει να εργαστούμε σκληρά επ' αυτού. Νομίζω ότι αυτό που είπα για τους άλλους ευάλωτους πληθυσμούς ισχύει και για τους ανθρώπους ε, με διαφορετική καταγωγή. Σίγουρα θα παλέψω, θα ε, δράσω ενεργά για να διασφαλίσω και να εφαρμόσω την αρχή της έλλειψης διακρίσεων. Για οποιοδήποτε λόγο δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή των μη διακρίσεων. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη αλλά και από τις εταιρείες. Πολλές έξυπνες εταιρείες έχουν αρχίσει να κατανοούν ότι η διαφορετικότητα αποτελεί τεράστιο ε, στοιχείο θετικό για αυτές. Ας ε, τις ενισχύσουμε και ας το πάρουμε ως καλό παράδειγμα. Κύριε Πάτεν. Δεν ε, το χάφτω αυτό κύριε ε, Σμιτ. 20 χρόνια ε, μετά από όλη αυτή την νομοθεσία κατά των διακρίσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και συνεχίζει να κάνει διακρίσεις με βάση το χρώμα. Οι ίσες ευκαιρίε και η πρόσβαση ανεξάρτητα από την καταγωγή και την εθνότητα είναι κάτι για το οποίο έχετε υποσχεθεί ξεκάθαρες δράσεις. Όμως δεν έχετε τίποτα να πείτε, ούτε καν ότι είστε ε, εντάξει ε, για τα του οίκου σας. Γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε ε, άμεσα, τουλάχιστον στο δικό σας τμήμα. Θα το κάνετε. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω πραγματικά και δώστε μου την ευκαιρία. Δεν έχω γίνει καν επίτροπος ακόμα, είμαι μόλις υποψήφιος αλλά η έλλειψη διακρίσεων είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξή μας ε, και είναι και στην ημερήσια διάταξη ολόκληρης της Επιτροπής, ειδικά της ε, εκλεγμένης Πρόεδρου. Ε, πραγματικά, δεν είναι όμως εύκολο. Είναι εύκολο να δακτυλοδεικτείς, να κατηγορείς, αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις εντάξει, 20 χρόνια είναι το παρελθόν, θα δούμε το μέλλον. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο για το παρελθόν, μπορεί να είμαι υπεύθυνο για το μέλλον. Θα έρθω εδώ σε 5 χρόνια και τότε μπορείτε να αξιολογήσετε την κατάσταση. Κύριε Πιθάρο. Πισάρο, συγγνώμη. pela profundidade das suas respostas. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας μέχρι τώρα. Παρά κάποιες θετικές εκκλήσεις το 2017, εξακολουθεί να υπάρχουν 113 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό για την ομάδα μας, τους σοσιαλιστές, είναι εντελώ απαράδεκτο. Γι' αυτό σας ρωτώ, κύριε Υποψήφια Επίτροπε, δεσμεύεστε να υποβάλλετε μια στρατηγική, να παρουσιάσετε μάλλον μια στρατηγική ε, καταπολέμησης της που θα καλύπτει ε, που θα είναι γενική και ολοκληρωμένη και θα ε, προλαβαίνει την ε, φτώχεια για τους εργαζόμενους, τις ανισότητες στους μισθούς, την έλλειψη της στέγασης σε προσιτές τιμές και την απασχόληση των νέων. Ειδικά για τους χρόνια άνεργους τα ποσοστά είναι πολύ ψηλά και παραμένουν ψηλά. We um, Σας ευχαριστώ. Έχουμε φιλόδοξους στόχους. 20 εκατομμύρια λιγότεροι άνεργοι. Αλλά δεν το πετύχαμε το στόχο αυτό. Υπήρξαν βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο που είχαμε θέσει το 2010. Πιστεύω πως ε, γίνεται πολύς λόγος για την ε, φτώχεια και είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι στο πλουσιότερο μέρος του κόσμου υπάρχουν τόσοι πολλοί, ένα στους πέντε που ζουν στη φτώχεια ε, και κάποιες φορές μάλιστα με μεγάλη φτώχεια. Χρειάζεται αποτελεσματική πόρη χρηματοδότηση για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση. Χρειάζεται και μια καλή στρατηγική για να το καταφέρουμε αυτό. Και ε, είναι προς το συμφέρον όλων. Κάθε κράτος μέλος και της Ένωσης της ίδιας Πρέπει δηλαδή πρώτα να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Υπάρχει αυτή η ιδέα ότι τουλάχιστον 25% το Κοινοβούλιο προτείνει περισσότερο ε, ότι τα κονδύλια που πάνε για ε, ένταξη να πάνε για την καταπολέμηση της στόχιας. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της στόχιας. Τα παιδιά τα συζητήσαμε, είναι πολύ σημαντικά ε, τα παιδιά για την καταπολέμηση της στόχιας και η εγγύηση για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά για την καταπολέμηση της στόχιας και εντάσσεται στη γενική στρατηγική. Νέοι, μάλιστα νέοι, πολύ συχνά δεν είναι καλά καταρτισμένοι, χρειάζεται να ε, καταρτιστούν. Μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους, ε, ε, ανθρώπους με, ίσως με αναπηρίες που δεν βρίσκουν δουλειά. Και μόνοι γονείς. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι, κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν στη φτώχεια. Ε, πρέπει λοιπόν, αυτό το έχουμε ήδη αποφασίσει, ε, να βρούμε γραμμές ε, και για τις ε, συστάσεις αναχώρα για να εστιάσουμε. Γιατί και εδώ δεν υπάρχει μία ομοιόμορφη προσέγγιση. Πρέπει να δούμε τις χώρες, τις περιφέρειες, την αστική φτώχεια, την, την φτώχεια της υπαίθρου ε, και ούτω καθεξής, γιατί τελικά εκεί το κράτος μέλος θα πρέπει να παίξει επίσης σημαντικό ρόλο. Μάλιστα, κύριε Πισάρο, ρώτησε κύριε Σμιτ, για να καταπολεμήσουμε την ένδυα θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα του μήνυμου μισοδήματο. και θα πρέπει να οφείλω να σας ρωτήσω αν είστε προσιλωμένος σε μια νέα ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για αξιοπρεπή μήνυμου εισοδήματα που θα θεσπίζουν μήνυμου στάνταρ για τα εθνικά συστήματα ώστε να προβλέπετε κοινωνική ε, για όλ, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να δεσμευτώ για το είδος του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να είναι οδηγία, μπορεί να είναι ένα άλλο πλαίσιο. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να έχουμε το σωστό επίπεδο ελάχιστου εισοδήματος που είναι όμως απαραίτητο. Και το είπα και προηγουμένως, ότι είναι απαραίτητο μέσο, διότι Γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα στις κοινωνίες μας. Δεν θα, σας, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, όμως είναι κομμάτι μιας γενικής στρατηγικής. Απασχόληση, δεξιότητες, εκπαίδευση, στέγαση. Στέγαση είναι σημαντική αν θέλουμε πραγματικά να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Αν ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σε ένα σωστό σπίτι, σε ένα αξιοπρεπέ σπίτι, δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τη φτώχεια και ούτε και να βρει δουλειά. Και είναι ένας φαύλος κύκλος που πρέπει εμείς να τον σπάσουμε. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνεχίζω μια προηγούμενη ερώτηση για τον ρόλο που θα πρέπει όλοι να παίξουμε στην υποστήριξη των πολιτών και της ε, ψυχικής υγείας τους. Πολλοί μας ε, βλέπουν και μας ακούν και ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα ψυχικής υγείας πάνω από το 4% είναι το κόστος αυτό το, ως προς το ΑΕΠ. Και έχουν και χαμηλότερη απασχόληση οι άνθρωποι αυτοί με ψυχικά προβλήματα. Θα έχουμε τις σωστές πολιτικές. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για όλα τα εκατομμύρια των πολιτών που εκπροσωπούμε και τα τρία θεσμικά όργανα. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ειδικέ ε, δράσεις που προτίθεστε να αναλάβετε για την ψυχική υγεία. Ε, στον χώρο εργασίας. Αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική ε, ε, για άτομα με αναπηρίες. Και αυτό είναι ένα τμήμα της πολιτικής αυτής. Θα πρέπει να βρούμε κάποια προγράμματα για τους ανθρώπους αυτούς για να εργάζονται. Μπορεί να μπορούν να εργάζονται, αλλά δεν μπορούν να εργάζονται ενδεχομένω σε οποιαδήποτε δουλειά, με πλήρης ωράριο. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς εντάσσονται σε ένα χώρο εργασίας και σε μια θέση εργασίας. Οι εταιρείε που το κάνουν αυτό χρειάζονται πλαισίωση, χρειάζονται βοήθεια. Ε, είναι μια συνολική στρατηγική. Όταν ήμουν υπουργό ε, εργασία, συνεργάστηκα με τον Υπουργό Υγεία και Οικογένεια και Κοινωνικών Υποθέσεων για να βγάλουμε κάποιε κατευθυντήριες γραμμέ ένα οδηγό συμβουλών για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν αυτό το κίνδυνο αλλά και δεσμεύονται για να έχουν ισχυρή κοινωνική ε, παρουσία και ευθύνη. Για να ε, ε, προσλαμβάνουν ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η κοινωνική οικονομία είναι ένας τομέας που μπορεί να ασχοληθεί καλύτερα με αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το προωθήσουμε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να έχουν δυσκολίε ε, σε ορισμένες επιχειρήσεις, αλλά όταν είναι διαφορετικό το περιβάλλον, στην κοινωνική οικονομία τη λεγόμενη, ε, μπορεί να είναι και αυτό μια απάντηση. Ε, επερώτησε. Ψηφιοποίηση. Συχνά συγκρούεται με την οργάνωση και τα σχήματα εργασίας. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε burnout ε, τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Αναφερθήκατε σε αυτό. Θα είναι η προτεραιότητά σας η ανανέωση ε, των ε, προτάσεων και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψυχική υγεία. Κοιτάξτε, θα πρέπει να συνεργαστώ και με την αρμόδια επίτροπο για τα θέματα υγείας και να συντονιστούμε. Αλλά αυτό το θέμα δεν μπορούμε να το διακόψουμε εδώ, θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Και φυσικά ε, θα το κοιτάξω μαζί με την ε, αρμόδια επίτροπο για θέματα υγείας ε, θα έχουμε μια συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Ήδη ανέφερα προηγουμένως ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν αρχίσει συζητήσεις για θέματα ψυχικών νοσημάτων και ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας, όπως είναι το στρες και το burnout, στο οποίο αναφερθήκατε. Θα πρέπει να διευρύνουμε και τις γνώσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε αυτά να τα προλαμβάνουμε γιατί σε πολλά από τα ζητήματα αυτά, όταν έχει έρθει η ώρα της θεραπείας, είναι ήδη πολύ αργά. Αρκετά αργά, μας περιπτώσει, δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ αργά. Αλλά αυτό που χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική πρόληψη. Όταν αρχίζει ο κόσμο να έχει ένα πρόβλημα, όχι αφού έχει εγκατασταθεί απολύτω το πρόβλημα. Και αυτή η προληπτική πολιτική θα πρέπει να είναι ενταγμένη ε, στην όλη μα προσέγγιση για θέματα υγιεινής και ασφάλισης στην εργασία. Η κυρία Σαϊμπή, παρακαλώ. Καλημέρα, κύριε υποψήφια επίτροπε. Είμαι ικανοποιημένη που σας άκουσα να μιλάτε για το θέμα της ουμπεροποίησης της εργασίας που αγγίζει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη παγίδα. Περνάνε οι μισθωτοί ω αυτοαπασχολούμενοι για να μπορεί κανεί να αποφύγει τι κοινωνικέ υποχρεώσει. Έτσι λοιπόν για αυτούς ε, του ε, εργοδότε θα πρέπει να βρούμε τρόπο να τους ελέγξουμε και να τους επιβάλλουμε κυρώσει. Υπάρχουν τρία κριτήρια που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δούμε ακριβώς πώς είναι ένας μισθωτός. Αυτά τα κριτήρια δεν έχουν ε, διατηρηθεί ξεκάθαρα στην αντίστοιχη οδηγία που αναφέρατε. Ε, υπάρχουν αυτοί στις πλατφόρμες που μας λένε ότι η οδηγία είναι πολύ καλή, αλλά εμάς δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και υπάρχουν ε, αυτοί που μεταφέρουν ε, με το ποδήλατο, οι οδηγοί, αυτοί που είναι στο Μαδρί, στη Μαδρίτη, στις Βρυξέλλες, αυτοί λένε ότι δεν είναι εργαζόμενοι, ότι είναι εταίροι. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτοί θα αναγνωρίζονται ως μισθωτοί. Αναφέρατε τη, μία ε, κοινωνική διάσκεψη για το θέμα. Ποια είναι τα συμπεράσματα που θέλετε να βγουν. Ε, μπορείτε να δεσμευτείτε για την έγκριση μιας συγκεκριμένης ε, οδηγίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Και εγώ είδα αυτή την εκπομπή σε ένα γαλλικό κανάλι για την κατάσταση μια σειρά εργαζομένων στις πλατφόρμες. Πολύ ενδιαφέρουσα να σας πω ότι μου άνοιξε κάπως τα μάτια όσο δεν είχαν ανοίξει ήδη. Εγώ πραγματικά ε, μέσα στην επιστολή της αποστολής μου έχω αναφέρει ότι θα ασχοληθώ με τα άτομα που εργάζονται στις πλατφόρμες. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε πραγματικά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχουμε και την κρίση του δικαστηρίου αυτή τη στιγμή για τους όρους που πρέπει να πληρούνται ώστε κανείς ε, να μην θεωρείται αυτό αποσχολούμενος ή ανεξάρτητος αλλά μισθωτός και ε, θα πρέπει με βάση αυτά τα θεσπίσματα να ε, ορίσουμε ξεκάθαρα, έχουμε δηλαδή καθήκον να ορίσουμε ξεκάθαρα το καθεστώς του ανεξάρτητου εργαζόμενου, το αυτοαπασχολούμενου και να τον αντιπα αντιδιαστήλουμε ε, στον μισθωτό, με το μισθωτό. Αυτό ακριβώς ε, πρέπει να γίνει ε, προς όφελος των εργαζόμενων στις πλατφόρμες. Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω. Δεν θέλω απλώς μια διάσκεψη για αυτό το θέμα. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να παρακάμψεις, ε, το έδειξε και στο φιλμ αυτό, να παρακάμψεις τον ορισμό ή τους ορισμούς. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι ορισμοί, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρα θεσπισμένα δικαιώματα και λέω για όλους τους μισθωτούς. Είτε είναι ε, ανεξάρτητοι είτε πραγματικοί μισθωτοί Γιατί μόνο όταν όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, τότε θα μπορεί, μόνο τότε δεν θα μπορεί κανείς να παίζει με τις ε, λέξεις και τις έννοιες. Και θα έχουν οι άνθρωποι το καθεστώς που θέλουν και που πρέπει να έχουν. Επερώτηση, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Τώρα. Αναφέρεται ότι το ζήτημα αυτό είναι μια, ας πούμε, ε, ένα θέμα που ενδεχομένως ε, να έχουν και άλλοι επιτροποί στην αρμοδιότητά τους. Ε, η κυρία Φερστάγκερ έχει μια νέα οδηγία για τις ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνει τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες. Υπάρχει λοιπόν σύγκρουση ε, αρμοδιοτήτων. Τι, καταλαβαίνετε ποια είναι η ανασυχία μας. Εμείς δεν θέλουμε να δούμε μόνο τον ανταγωνισμό στην αγορά των υπηρεσιών. Κύριε Επίτροπε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος. Φοβάμαι να πάμε από μια ξεκάθαρη κοινωνική διάσταση, μια ξεκάθαρη πρωτοβουλία τέτοια ε, προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα μιλήσουμε πραγματικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες. Πραγματικά το είπα με την ε, δήλωση της αποστολής μου. Εγώ είμαι απλώς ένας ε, φτωχός επίτροπος που δεν έχει καμία επιρροή. Όχι. Δεν αφήνομαι έτσι ε, να παρετηθώ από τις ε, αρμοδιότητες και τα δικαιώματά μου. Άκουσα κι εγώ, και μάλλον διάβασα κι εγώ αυτά που είπε η κυρία Φεστάγκερ. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Είπε ότι θέλει μια ψηφιακή οικονομία στην υπηρεσία των πολιτών, των ανδρών και γυναικών. Και ε, πραγματικά πρόκειται για μια ξεκάθαρη δέσμευση. Όλοι έχουμε πιστεί από την Καλιφόρνια ως την Ευρώπη ότι δεν μπορούμε να κοιτάμε τη νέα ψηφιακή οικονομία μόνο υπό το πρίσμα της αγοράς, των επιχειρήσεων, της ανταγωνιστικότητας. Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στην ψηφιακή οικονομία δεν είναι τα μηχανήματα, είναι οι άνθρωποι το να φτιάξεις μια ψηφιακή οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο, αυτό είναι που θα ε, το επιθυμητό. Αυτό θα υπερασπιστώ και θα έχω και την κυρία Φερστάγκερ στο πλάι μου, η οποία ε, είναι ε, υπέρ αυτού του νέου μοντέλου που φαίνεται ότι παντού υπάρχει. Ο κύριος ευχαριστώ. Ε, εξ ονόματος των δημοκρατών, Θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία για μας είναι οι συνθήκες εργασίας. Ε, γι' αυτό υποστηρίζουμε ε, ένα κατώτατο εισόδημα αξιοπρεπές και υπάρχει ένας αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ένα άμκα ας πούμε για όλους τους πολίτες, να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική προστασία και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς αυτά δεν συμβαίνουν. Είπατε ήδη πολλά για την προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εσείς πώς θα εξασφαλίσετε δηλαδή τα δικαιώματά τους. Ποια είναι τα στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για σας. Πώς θα εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διαφάνεια στις πληρωμές και στην απόσπαση των εργαζομένων. Καταρχάς, το θέμα της κοινωνικής προστασίας. Είναι πραγματικά κομβικό. Και η έγκριση των συστάσεων για την κοινωνική προστασία είναι σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει και ένας μηχανισμός για το πώς τα κράτη-μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τις συστάσεις αυτές. Και θα πρέπει πραγματικά να οργανώσουμε μια συνέχεια, ένα follow-up για την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο αυτό. Θα πρέπει να εφαρμόζονται ε, με τρόπο αποτελεσματικό και δίκαιο αυτές οι συστάσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Για τη δεύτερη, θα πρέπει να σας παραπέμψω σε αυτά που είπα για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Εργασίας, Labor Authority. Ε, δημιουργήσαμε αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Εκεί συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι και οι κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τη λειτουργία ε, αυτής της αρχής. Αυτό θέλω το συντομότερο να αρχίσει να λειτουργεί. Είναι σημαντικό αυτό και για την απόσπαση. Ενδεχομένως δεν είναι σημαντικό στο μέλλον και για κάθε είδους θέματα που έχουν σχέση με τις εργασιακές υποθέσεις, ακόμα και ζητήματα ασφάλειας. Γιατί πολύ συχνά οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι δεν είναι εκείνοι που έχουν και την καλύτερη προστασία σε σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία τους. Αυτό πρέπει να το φροντίσουμε. Η εφαρμογή, η υλοποίηση. Το θέμα δεν είναι να νομοθετείς, είναι να υλοποιείς την νομοθεσία. Και εδώ τα κράτη-μέλη έχουν και αυτά την ευθύνη τους. Ε, με αυτά θα πρέπει να συζητούμε και να αδράξουμε την καλή ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με πολλές συστάσεις οι οποίες τώρα αφορούν τα κοινωνικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις συστάσεις αναχώρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση των κρατών μελών, να σέβονται τους κανόνες και να το καταλάβουν αυτό και να έχουν καλές πολιτικές σε όλα τα θέματα που μόλις αναφέρατε. Συμπληρωματική ερώτηση, επερώτηση. Μάλιστα. Και η επόμενη ερώτηση αφορά ε, τις ε, εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές. Το 1994 εγκρίθηκε μια οδηγία ε, για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι πολλές οι προκλήσεις από την οδηγία αυτή ακόμα και πολλά τα προβλήματα. Πώς θα φροντίσετε να υπάρξουν κυρώσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Και τι γίνεται με την υλοποίηση στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται καλύτερα οι ίδιοι εργαζόμενοι για τα δικαιώματά τους. Αυτή η οδηγία στην οποία αναφέρεστε αφορά τα επιχειρησιακά συμβούλια. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες σε αυτή την οδηγία. Ήταν τότε μεγάλη πρόοδος, αλλά έχει και αδυναμίες. Γιατί είναι μια λειτουργία που λειτουργεί έτσι κάπως ε, εθελοντικά. Και άρα ορισμένοι την εφαρμόζουν και άλλοι πάλι όχι. Και εκείνοι που εφαρμόζουν την οδηγία, καμιά φορά δεν την εφαρμόζουν ε, ουσιαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας Θα καλέσω τους κοινωνικούς εταίρους ε, στη διαβούλευση αυτή. Δεν είμαι υπεραισιόδοξος το ομολογώ. Αλλά είναι σημαντικό να το συζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Το έχουν ήδη συζητήσει. Αλλά πρέπει να αναλύσουν πραγματικά τις αδυναμίες, τις οδηγίες, τι μπορεί να βελτιωθεί. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι καλές, αλλά δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Γιατί αν αυξήσουμε τις κυρώσεις, ποια θα είναι η συνέπεια θα είναι ακόμα λιγότερες εκείνες οι εταιρείε που θα μπαίνουν στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Γιατί σου λέει δεν αναβάνω τον κίνδυνο να μου επιβληθούν κυρώσεις, οπότε δεν το υιοθετώ αυτό το μέτρο καθόλου. Θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική αξιολόγηση ποια είναι τα αποτελέσματα που έχει φέρει η οδηγία, γιατί υπάρχουν σίγουρα και θετικά, ποιες είναι οι αδυναμίες, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη εφαρμογή και πάλι της οδηγίας η Επιτροπή σας πρότεινε κάποια μέτρα και διάφορα απορρίφθηκαν βέβαια. Αυτό είναι στην ημερησία διαταξή μας, θα το κοιτάξουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω προς ποια κατεύθυνση θα καταλήξουμε. Είναι σημαντική όμως η οδηγία και θα πρέπει να τη λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Σπάρεντακ. Η κυρία Σπάρεντακ. Thank you. Um, in EU, e more people are homeless and... Ευχαριστώ. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άστοιχοι και πολλοί αγωνίζονται να βάλουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, μέσα στο πλαίσιο της ε, δέσμευσής σας για μείωση της ε, φτώχειας, ε, θα αναλάβετε την παροχή στέγασης. Που στη χώρα μου, πολλοί κόσμος δεν μπορεί να βρει κοινωνική στέγαση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εμποδίσει τη χώρα μου να κατασκευάσει και να δώσει προσφέρει κοινωνική στέγαση στους ε, άπορους. Ε, εσείς θα θελήσετε και θα στοχεύσετε ε, στην μετατροπή της ευρωπαϊκής πολιτικής ώστε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και να προσφερθεί στέγαση. Μάλιστα, ξέρετε και εγώ προέρχομαι από μια χώρα που υπάρχει θέμα στέγασης, θέμα οικιστικό, το οποίο υπάρχει σε πολλές χώρες μέλη. Αν και η αρμοδιότητες ε, είναι των κρατών μελών σε αυτό το τομέα, πιστεύω πως η Ένωση ε, μπορεί να παίξει έναν ε, ρόλο προώθησης ενθαρρύνοντας καταρχάς περισσότερες επενδύσεις στην στέγαση και τώρα έχουμε σκοπό να φτιάξουμε νέα επενδυτικά εργαλεία. Όταν μιλάμε για ένδια, η επένδυση στη στέγαση είναι ακριβώς ένα εργαλείο για να μειωθεί η ε, να μειωθούν οι άστεγοι οι άποροι, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ε, στέγη δεν βγαίνουν εύκολα από την κατάσταση φτώχειας. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη για την κοινωνική στέγη υπό δίκαιους όρους, και με αναφέρατε το θέμα του ανταγωνισμού. Πρέπει πράγματι αυτό να το αναλύσουμε και να δούμε ακριβώς αν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες αυτές ανταποκρίνονται στην κατάσταση, στην πραγματικότητα επιτόπου, αλλά υπάρχει ανάγκη για προώθηση των επενδύσεων στην στέγαση σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Ε, όχι, και βέβαια μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των κρατών το, της Ένωσης, με θα προσπαθήσω να εντάξω αυτή τη διάσταση στον αγώνα για την καταπολέμηση της φτώχειας και να περιλάβω την δέσμευσή μας για ένταξη. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για αυτή σας την απάντηση, αλλά θα αναλάβετε δραστήρια αυτή την ευθύνη για ευρωπαϊκή στρατηγική για την κοινωνική στέγη, γιατί είπατε πως ε, θα βοηθήσετε τους νέους να έχουν δίκαιη πρόσβαση στην ε, αγορά, αλλά θα πρέπει να δεχτείτε ότι για τους νέους είναι το ίδιο σημαντικό και η πρόσβαση στην ε, στέγη. Μάλιστα δεν είναι μόνο ο Επίτροπο για την Απασχόληση και Κοινωνικέ Υποθέσει μπορεί να το κάνει αυτό μόνο. Στον οικονομικό θέμα πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλου επιτρόπου. Είναι οικονομικό, ε, ε, δημοσιονομικό θέμα να δούμε τι είδου μέσα μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να ενθαρρύνουμε τι επενδύσει στην ε, στέγαση. Είμαι κομμάτι μια ομάδα. Δεν είμαι ένα που αποφασίζει ε, τι θα κάνει μόνος του. Η Επιτροπή είναι ομάδα ε, και ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι στόχος αυτής της Επιτροπής να κάνει κάτι για την κοινωνική στέγη και το οικιστικό πρόβλημα σε πολλά μέρη της Ευρώπης που συνδέεται με τους νέους, με τα παιδιά, με τις θέσεις απασχόλησης. αν δεν έχεις στέγη δεν μπορείς εύκολα να βρεις και δουλειά. Θα, εγώ θα πιέσω λοιπόν για την εξέβρεση λύσεων δεδομένων στις περιορισμένες αρμοδιότητες που έχει η Ένωση και λαμβάνοντας υπόψη ε, τι ε, οικονομικά μέσα που μπορούμε να κινητοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα σε αυτό το πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο τομέα. Ο κύριος Κάνιας estamos de acuerdo que esta ser Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ο κοινωνικός πυλώνας ε, των δικαιωμάτων για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να φτάσουμε στους στόχους μιας Ευρώπης ε, των πολιτών και για τους πολίτες της. Εκεί συμφωνούμε όλοι. Ποια είναι λοιπόν η κοινωνική οικονομία και ο ρόλος της. Είναι θεμελιώδης τρία εκατομμύρια επιχειρήσεις ε, που ε, εργοδοτούν ε, περίπου 14 εκατομμύρια πολίτες και παράγουν το 8% του ΑΕΠ. Οι κοινωνικές αυτές επιχειρήσεις και δομές για την οικονομική, κοινωνική συνοχή, την εδαφική είναι ένα μοντέλο βιώσιμο που δουλεύει με τους πιο ευάλωτους και αυτό το αναγνωρίζουν μόνο ορισμένα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο με διάφορες νομικές ε, μορφές. Θα καταθέσετε μια πρόταση για να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο και ομοιογενές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική οικονομία κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Απάντηση. Να σας καθησυχάσω, είμαι μέγας υποστηρικτής κοινωνικής οικονομίας. Έχω διατελέσει και υπουργό κοινωνικής οικονομίας. Πιστεύω στο σημαντικό πρωταγωνιστικό της ρόλο ήδη από τώρα. Και σίγουρα έχει ακόμα δυναμικό να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία. Ιδιαίτερα δεδομένων των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, η φτώχεια, αποκλεισμό, όλα αυτά τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα καμιά φορά αν έχουμε ισχυρή κοινωνική οικονομία. Σίγουρα το μοντέλο τη κοινωνική οικονομία δεν είναι το ίδιο σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να σεβόμαστε και τι διάφορε κουλτούρε και παραδόσεις. Το ίδιο ισχύει και για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Πρέπει να σεβόμαστε ε, τα διαφορετικά μοντέλα που υπάρχουν στι διάφορε χώρε. Ε, εκεί όμω χωράει ακόμα πολύ δράση, κοινή δράση. Και το 2011 ο Επίτροπος Μπαγνιέ και ο Επίτροπος Άντορα, αν δεν θυμάμαι, και τα Γιάννη τότε, είχαν ε, μια διάσκεψη για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που δημιούργησε πραγματικά μια θετική ε, δυναμική. Ε, έχω λοιπόν την ιδέα μαζί με άλλους επιτρόπους και πάλι, δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα και ευθύνη. Μαζί με άλλους επιτρόπους να επαναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία να φέρουμε τους ενδιαφερομένους εδώ και να έχουμε ένα σχέδιο για την πρόθεση της κοινωνικής οικονομίας σε σχέση και πάντα με τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε στις κοινωνίες μας και να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο της κοινωνικής οικονομίας. Προηγουμένως ανέφερα τα οικονομικά, ε, να προωθήσουμε και τα οικονομικά και τα θέματα θέσεων εργασίας. Υπάρχει δυναμικό εκεί, πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Η εσωτερική αγορά είναι σημαντικό. Η κοινωνική οικονομία θα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα στην εσωτερική αγορά με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Πραγματικά προσβλέπω στη συνεργασία με άλλους επιτρόπους στην κατεύθυνση αυτή, έτσι ώστε η κοινωνική οικονομία να γίνει ακόμα πιο στιβαρή και να εδρεωθεί στην Ευρώπη και να είναι τμήμα και στοιχείο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Και αυτό συνδέεται και με την κοινωνική εταιρική ευθύνη που αναφέρατε εσείς κύριε Κιμπουρόπουλη. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Συγκεκριμένα ρωτάω όμως. Ε, θα ήταν απαραίτητο να έχουμε ένα ομοιογενές πλαίσιο με σαφείς κανόνες, χειροπιαστές καταστάσεις. Υπάρχουν προκλήσεις και σε αυτή τη θητεία και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε όπως είναι ε, η αντασφάλιση του επιδόματος ανεργίας. Η νεανική ανεργία είναι τραγική σε κάποιες χώρες, με απαράδεκτα ποσοστά που θα πρέπει όλοι να καταπολεμήσουμε. Και έχω μια ερώτηση σχετική. Θα υποστηρίξετε το 10% αυτό το υποχρεωτικό ε, αποθεματικό για την εργασία των νέων και για χώρες που πλήγονται περισσότερο, που πλήττονται. Μήπως σκέφτεστε και το 15% γιατί είναι πραγματικά μάστιγα, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Ε, θα πρέπει αυτή η θητεία να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Σύντομη απάντηση. Εάν θέλουμε να εναρμονίσουμε πραγματικά το καθεστώς αυτό που ονομάζουμε κοινωνική οικονομία που στη Γερμανία πούμε, το λένε τελείω διαφορετικό. Στη Γερμανία η κοινωνική οικονομία δεν καταλαβαίνουν τι είναι, να το πει έτσι. Αλλά έχουν ένα τέτοιο κλάδο πάρα πολύ ισχυρό. Αν θέλουμε να το εναρμονίσουμε δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Μπορούμε να έχουμε μια πολύ πραγματιστική, ρεαλιστική προσέγγιση και να δημιουργήσουμε κοινού κανόνε παιχνιδιού για όλου για τις ενώσεις, τα σωματεία, τις επιχειρήσεις που θεωρούν ότι ανήκουν στον κοινωνικό τομέα της αγοράς. Συμπροματικό. Α, για τη δεύτερη ερώτηση τώρα. Πολύ σημαντική αυτή η νεανική ενεργεία. Και αυτό είναι και παραμένει προτεραιότητα απόλυτη στο θεματολόγιο μας. Τώρα δεν θέλω να σας δώσω ε, ε, ε, απάντηση με στοιχεία 3% ή 15%. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, καλύτερα, να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα μέσα. Μιλήσαμε πολύ για την εγγύηση, για την νεολαία. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η επαιδεία, η κατάρτιση. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και φυσικά οι πόροι που έχουμε για την νεολαία για την εγγύηση, για την αλλαγή, για την νεανική ανεργία θα πρέπει να δοθούν εκεί που είναι και παραμένει πρόβλημα. Εκεί που είναι πολύ χαμηλή η νεανική ανεργία μπορούν μόνοι τους να το λύσουν. Αλλά εκεί που υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ενεργείας των νέων θα πρέπει να εστιάσουμε τους πόρους μας. Ο κύριος Χέτμαν, τελευταία ερώτηση για σήμερα. Και όλες, λέει ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλήσατε ε, μακροσκελώς ε, για την απόσπαση των εργαζομένων. Ήθελα όμως ε, να σας κάνω μια πολύ απλή και σύντομη ερώτηση. Οι διευθυντές επιτρέπουν την δημοσίευση μόνο σε μία ιστοσελίδα για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την απόσπαση. Αυτό λένε οι οδηγίες. Όμως, δυστυχώς, δεν υπάρχει αρκετή πληροφόρηση. Τι βήματα θα κάνετε ώστε αυτές οι ιστοσελίδες πραγματικά να αντικατοπτρίζουν την πραγματική νομική κατάσταση στις χώρες που βλέπουμε αποσπασμένους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. It's again question of implementation. Πάλι είναι θέμα εφαρμογής. Δεν αρκεί να έχεις καλούς κανόνες, κανονισμούς, Πρέπει να διασφαλίζεις ότι αυτά που αποφάσεις πρέπει και να εφαρμόζονται. Να πω, να παραδεχτώ ότι αυτό δεν το ήξερα. Θα ελέγξω αν όντω ισχύει, αν όντω δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, αν οι ιστοσελίδες δεν είναι πλήρεις, αν τα στοιχεία που πρέπει να δοθούν δεν έχουν παραδοθεί. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν υφίσταται αυτό, θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη σωστή πληροφόρηση. Ξέρετε, ε, η απόσπαση είναι κάτι θετικό. Την παρουσιάζουμε σαν το ύψιστο κακό, όμως ε, ε, μπορεί να είναι κάτι θετικό όταν γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες. Θετικό και για τη χώρα και για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο Ακριβώς. Το, για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον όλες τις πληροφορίες για τους όρους. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Αν λοιπόν όντω ισχύει αυτό που είπατε, αν δεν δίνονται τα, οι πληροφορίες στο ίντερνετ, η Κομισιόν σίγουρα θα κάνει κάτι γι' αυτό και θα φροντίσει να ε, γίνει κάτι τέτοιο. Να παραδεχτώ όμως ότι δεν το ήξερα και πρέπει να το ελέγξω. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχω πάρει τη δουλειά, οπότε δώστε μου ε, έτσι ένα περιθώριο. Επερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να κάνω την τελευταία από όλε τις ερωτήσεις. Όταν μιλάμε για την εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων, τίθεται το εξή ερώτημα. Τι θα κάνετε με το δυσανάλογο διοικητικό φόρτο που επομίζονται κάποια κράτη-μέλη. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα είναι δίκαιη η μεταφορά εργαζομένων και υπηρεσιών και δίκαιη μέσα στα πλαίσια της οδηγίας. Νομίζω ότι εν μέρη ήδη απάντησα σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο και που κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί. Γιατί κάθε φορά όταν έχεις διοικητικό φόρτο, έχεις και κάποιες δεύτερες σκέψεις. Αναρωτιέσαι κατά πόσο χρειάζεται. Δεν θέλουμε τέτοιες σκέψεις. Θέλουμε κάτι το οποίο να θεωρείται απαραίτητο. Όχι κάτι που να κάνει δύσκολη τη ζωή των διοικητικών υπαλλήλων, των εργαζομένων, των χωρών που δέχονται ή που στέλνουν εργαζόμενους. Άρα θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που κάνει δίκαιη και αποτελεσματική την απόσπαση εργαζομένων. Ποια είναι τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. Πώς θα παρασχεθούν αυτά τα στοιχεία. Τι γίνεται αν δεν γίνει το περίφημο Α1 πριν από την απόσπαση. Τι γίνεται όταν γίνει λίγο μετά. Όλα αυτά είναι πρακτικά ζητήματα. Πρέπει να τα αξιολογήσουμε. Και με βάση την αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προσαρμογές, αν χρειάζονται φυσικά. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα καθιστά αδύνατη την απόσπαση. Μα έχουμε κάνει ένα σύστημα που, το κάνει, που την κάνει επωφελή για όλους. Ένα σύστημα που είναι προσβάσιμο σε όλους, γιατί υπάρχουν κανόνες Χωρίς κανόνες υπάρχει απόρριψη. Η απόσπαση είναι κομμάτι της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και ελεύθερης κυκλοφορίας. Πρέπει λοιπόν να γίνεται σωστά και δίκαια. Αυτό θα κάνουμε και σε επίπεδο διοικητικών διεργασιών. Ευχαριστώ. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα τα, τα πήρετε μπόνους κύριε Σμίτη. Δεν χρησιμοποίησα το σφυράκι μου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ερωτήσεις σας και για τις απαντήσεις σας. Και τώρα θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία ε, να κάνετε μια τελική ε, δήλωση για πέντε μόνο λεπτά. Σας ευχαριστώ, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ε, πολύ ενδιαφέρουσα επικοδομητική και κρίσιμη συζήτηση που είχαμε. Θα πρέπει να πω ότι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και ότι τα κράτη-μέλη και όλοι ερχόμαστε από τα κράτη-μέλη μας και έχουμε ευθύνε και δεν ξέρω και πολλά κράτη-μέλη που να γίνεται κάτι τέτοιο. Πραγματικά θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για το δημοκρατικό μας σύστημα και συγχαίρω το κοινοβούλιο μας, γιατί είμαι ακόμα μέλος του κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου μας που ε, εισήγαγε αυτή τη συζήτηση, αυτή την ανταλλαγή. Γιατί η δουλειά του Επιτρόπου θα πρέπει πολύ άμεσα να σχετίζεται με τη δουλειά εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, δεν είμαστε δεν μπορούμε να είμαστε μακριά από τα όσα συμβαίνουν εδώ. Συχνά ακούω ότι ναι, αυτοί οι επίτροποι δεν εκλέγονται κτλ. Ναι, αλλά εγώ έγινα υπουργό, α πούμε, χωρί να έχω εκλεγεί στο κράτο μέλο μου. Τώρα έχω εκλεγεί στο κοινοβούλιο και θα κρυθώ από εσά. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε κανένα νομίζω κράτος μέλος μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πολύ καταπληκτική ε, ιστορία. Μου άρεσε πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι πέφερα, αλλά ήταν σκληρή η ε, συνέντευξη και έπρεπε να είναι και σκληρή. Now, it's not because we had a good... Δεν είναι ότι επειδή κάναμε τώρα μια καλή συζήτηση σήμερα πως δεν θα πρέπει να έχουμε πολύ συχνά τέτοιου είδους συζητήσεις και θα επανέλθω οποτεδήποτε μου το ζητήσετε, οποτεδήποτε έχω την αίσθηση ότι πρέπει να σας μιλήσω, να πάρω τη γνώμη σας, να ακούσω τη γνώμη σας που θα είναι ίσως κάποιες φορές διαφορετική, επικριτική, αλλά νομίζω πως αυτό είναι που κάνει την ευρωπαϊκή πολιτική τόσο ζωντανή και δημοκρατική. Και γι' αυτό θα ήθελα να ε, πω ότι θα είμαι μαζί σας όσο γίνεται συχνότερα και θα συνεχίσω αυτό που, ε, ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε ένα μεγάλο κοινό project. Ε, παντού όλοι ο καθένας με βάση τα ιδανικά του και τις ιδέες του. Δεν είμαστε ίδιοι γιατί διαφορετικά θα ήταν μόνο ένα κόμμα εδώ πέρα που σίγουρα δεν θα το θέλαμε αυτό να συμβεί. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να υπηρετήσουμε τους λαούς μας, να υπηρετήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, να φέρουμε την Ευρώπη πάλι κοντά στον πολίτη. Και οι πολίτες μας έχουν την καθημερινή τους ζωή, έχουν τα καθημερινά τους προβλήματα και πρέπει εμείς να ασχοληθούμε με αυτά και με τα όσα ρωτάνε για τους ελάχιστους μισθούς, για τη φτώχεια, για τα παιδιά, για τα καθημερινά που απασχολούν τους συμπολίτε μας. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε να εξασφαλίσουμε πως οι οι πολιτικές μας εξυπηρετούν τους πολίτες μας στην καθημερινή του ζωή. Ότι μετά από πέντε χρόνια αυτή τη επιτροπή οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να πούν αν υπήρξε πραγματική θετική ε, πρόοδος, ότι υπήρξε κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ζωή μου μας, χάρη στην Ευρώπη. Ε, αυτή είναι η πρόκληση. Δεν είναι μόνο η ειρήνη, που η ειρήνη φυσικά είναι ένα πολύ σπουδαίο και σημαντικό θέμα, αλλά είναι η κοινή ευημερία, η ιδέα ότι όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι μέρη της κοινωνίας και να έχουν τις ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι που κάνει την Ευρώπη σπουδαία και πρέπει να υπερασπίσουμε αυτές τις αξίες, όχι μόνο με τα λόγια βεβαίως, συμφωνώ, αλλά καθημερινά με τις πολιτικές μας ενέργειες. αυτό οφείλουμε να κάνουμε από κοινού η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο βεβαίως, αλλά και αυτό μαζί με το Κοινοβούλιο, γιατί εσείς είστε η φωνή των συμπολιτών μας και πρέπει να ακούσουμε αυτή τη φωνή. Σας ευχαριστώ. Thank you uh, Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ως πρόεδρος με τη σειρά μου θα ήθελα να σχολιάσω μερικά πράγματα για να κάνω μερικά σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, για μένα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση, καθώς ήταν και η πρώτη μου. Και εσάς η πρώτη σας. Έχουμε κάτι κοινό, λοιπόν. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ε, για μένα η ευκαιρία που είχα να παρακολουθήσω τις ερωτήσεις σας που ήταν σκληρές και επικριτικές και πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Η κοινωνική διάσταση του χαρτοφυλακίου σήμερα ήταν πολύ πιο ζωντανή. Αυτό κυριάρχησε και λιγότερο η δημιουργία θέσεων εργασίας που βασικά είναι το κύριο θέμα του χαρτοφυλακίου του κύριου Σμιτ. Όταν μιλούμε όμως για την κοινωνική ένταξη των κοινωνικών αποκλεισμένων ε, ατόμων ας πούμε, που ανήκουν σε μειονότητες ή ατόμων με αναπηρίες, ε, δεν φαντάζομαι καλύτερη ένταξη στην κοινωνία από εκείνη μέσω της αγοράς εργασίας. Σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν πιστεύω, να δημιουργούμε βιώσιμες θέσεις εργασίας για εκείνους που τις χρειάζονται πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή αποκλείονται ε, σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολυτέλεια, γιατί υπάρχει τεράστια αναντιστοιχεία και χάσμα στην αγορά εργασίας. Τους χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους για να καλύψουμε το χάσμα και το έλλειμμα. Ε, επίσης, εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που είπατε κύριε Σμιτ σχετικά με τη συζήτηση ε, για τις βάσεις δεδομένων, για τον αντίκτυπο των πολιτικών μας και τις μελέτες αντικτύπου. Γιατί ε, ακούμε για την Κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση για χρόνια ολόκληρα. Και η αλήθεια ποια είναι. Το 1 τέταρτο των παιδιών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν στη φτώχεια. Στους δρόμους μας έχουμε 70% περισσότερους αστέγους από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία πρέπει να βασίζεστε. Λοιπόν, κάτι πάει στραβά ή δεν πάει τόσο καλά όσο φανταζόμαστε. Ε, το τελευταίο. Αυτό που ακούσαμε ήταν ένα πάρα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Θέλετε να ανοίξετε πάρα πολλά θέματα που αυτή τη στιγμή διχάζουν τα κράτη-μέλη αντί να τα ενώνουν. Γιατί θέλει να θέλετε να ανοίξετε πολύ ευαίσθητα κεφάλαια. Και το τελευταίο είναι ότι θα πρέπει να υποσχόμαστε μόνο αυτό που μπορούμε να εκπληρώσουμε. Γιατί οι προσδοκίες και ελπίδες των πολιτών είναι τεράστιες. Και υπάρχει και ένα τεράστιο κύμα ε, λαϊκισμού μεταξύ των πολιτικών σε διάφορα κράτη-μέλη, σε όλα βασικά. Άρα, κάποια από τα σχέδια που έχετε μπορεί να τύχουν ε, εκμετάλλευσης και κατάχρησης εάν δεν κάνουμε όλα αυτά που υποσχεθήκαμε. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα εσάς κύριε Σμιτ. Um, λοιπόν, πριν ε, κηρύξω το πέρα τη συνεδρίαση. Θέλω να σα πω ότι θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ και κλεισμένων των θυρών για να αξιολογήσουν την ακρόαση. Αμέσω μετά στι 12.30 δηλαδή με 1.30 στην αίθουσα ASP 1Ε2. ASP 1Ε2. Και επίση θα σας ζητήσω να κάνετε όλοι λίγη υπομονή γιατί δεν πρόκειται να είναι εύκολο η διαδικασία αξιολόγησης και η επιστολή αξιολόγησης είναι ε, απόρριτα. Δεν θα στείλουμε τίποτα με mail, όλα και κλεισμένο των θυρών μεταξύ των συντονιστών. Και η διάσκεψη των προέδρων θα ανακοινώσει ε, τα αποτελέσματα και τα δικά μας αφού ολοκληρωθούν όλες οι ακροάσεις. Λήξη συνεδρίασης.